κατιούσα πορεία από το περιθώριο 1,6 σε 125 εκατομμύρια. Δηλαδή, εάν λάβουμε υπόψη τις αρχικές προβολές και προβλέψεις, μιλούσαμε για 122 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά ότι οι προβολές αυτές των υποχρεώσεων για τη γεωργία γνωρίζουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή, ως προς αρχικές προβολές μέχρι το πρώτο προσχέδιο προϋπολογισμού που υπογράφεται από την Κομισιόν τον Απρίλιο μέχρι την τελική έκδοση η οποία αλλάζει άρδιν από αυτή την πλευρά από το amending letter του φθινοπόρου. Άρα μιλάμε για αύξηση 3,4% που είναι χαμηλότερο περιθώριο σε σχέση με τον ε, προϋπολογισμό του 2011 και ίσως αλλάξει κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας προτείνω σήμερα και γι' αυτό έρχομαι σε επαφή με όλες τις εξειδικευμένες επιτροπές είναι μια στρατηγική προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλεται. Δηλαδή, εξ αρχής θα ήθελα να ορίσετε τις προτεραιότητες που θεωρούμε ή θεωρείται ύψης της σημασίας για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2012. Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής λοιπόν 2020 και στα πλαίσια αρμοδιοτήτων αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογήσετε τις δικές σας προτεραιότητες για τον προπολογισμό του 2012. Να δείτε δηλαδή πού θα πρέπει να ενισχύσουμε την πλαισίωση και πού θα πρέπει να δοθεί μια νέα διάσταση, που υπάρχουν ειδικοί προγραμματισμοί και, όπου, και πού τα προγράμματα δράσης δεν απέδωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που δεν επαρκούν ή να δούμε που δεν απορροφήθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αφορά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τις πιλωτικές, διότι πρόκειται για προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα περιθώρια. Να δούμε δηλαδή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα περιθώρια και που είναι πιο περιορισμένα. Θέλουμε να έχουμε ένα προσχέδιο των πιλωτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων που θα εγκριθούν για το 2012 και η υπόδειξή μου θα ήταν να αξιολογήσουμε τα προγράμματα δράσης που ισχύουν ήδη, που είναι ενισχύ πριν εισαγάγουμε καινούργια θέματα ή δράσεις και να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς τους για να αξιολογήσουμε καλύτερα του, τους πόρους και να δούμε πού αποδίδουν. Άρα, θα πρέπει στη διαδικασία προϋπολογισμού να συμμετάσχουμε όλοι πέρα από τις ε, πολιτικές διαστάσεις της, Επιτροπής, ε, της εργασίας της Επιτροπής Προϋπολογισμών και να ορίσουμε τις προτεραιότητες που κάθε επιτροπή ορίζει και γνωρίζει πολύ καλύτερα. Και αυτό αφορά ολόκληρη τη διαδικασία, γιατί δεν σημαίνει ότι εκτιμούμε καλύτερα την Επιτροπή στις προτάσεις της 20 Απριλίου, αλλά θα προετοιμάσουμε και τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για να έχουμε το δημοσιονομικό μας έγγραφο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα πλαίσια του ίδιου του προϋπολογισμού. Άρα εσείς έχετε το λόγο γιατί φέρετε μεγάλη ευθύνη και πρέπει να είσαστε αποδοτικοί και συνεκτικοί στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Ευχαριστούμε τη Φραντσέσκα come sta impostando il lavoro in Commissione e Θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ορίσουμε μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ τις προτερότητες όλων των πολιτών. Και τώρα ο, το λόγο έχει ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλτζάνη. Ε, εργαστήκαμε πολύ καλά και πέρσι και φέτος είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μία καλή διάρθρωση της συζήτησης. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πρόκειται για μία συζήτηση η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε για ορισμένες ε, γενικές αρχές. Τα περιθώρια είναι περιορισμένα και μιλάμε για τέσσερις βασικές συνιστώσεις του προπολογισμού για τη γεωργία. Μιλάμε για τις άμεσες πληρωμές, τα μέτρα υπέρ της αγοράς, ε, την αγροτική ανάπτυξη και τα εξειδικευμένα προγράμματα. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων δεν είναι ξισορροπημένες και υπάρχει μεγάλη ανελιξία ιδιαίτερα ως προς τις άμεσες πληρωμές. Σε σχέση με τα μέτρα υπέρ της αγοράς, εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ, διότι μας ενδιαφέρουν ε, οι προσδοκίες. Υπάρχει μεγάλη ε, δυσανεξία στην αγορά αγαθών, στην αγορά των commodities Υπάρχουν τομείς που γνωρίζουν μεγάλη κρίση, δηλαδή του χειρίου κρέατος, του βοήου κρέατος και γνωρίζοντας και τους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε σχέση με τις διατροφικές ανάγκες. Μιλώ για την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική, στην τραγωδία της Ιαπωνίας και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν από αυτές τις ε, δυσίωνες καταστάσεις. Για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καλύψουμε τις διατροφικές μας ανάγκες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα χρηματοοικονομικά μέσα μέσα στα πλαίσια του 2011 2012 για να ορίσουμε τις δυσκολίες σε σχέση με τα ειδικά προβλήματα, πέρα από το γεγονός ότι οι εγγραφές είναι περιορισμένες. Καθίσταται σαφές ότι η Επιτροπή Γεωργίας θα ταχθεί υπέρ των πιο ευάλωτων ε, κατηγοριών. Επίσης θα γίνεται διανομή φρούτων στα σχολεία για να καταπολεμήσουμε την παχύσαρκία και επίσης θα υπάρχει παροχή ε, γάλακτος στα σχολεία, όπως είχαμε ορίσει και πέρσι. αυτά τα μέτρα, σε αυτά τα μέτρα θα δοθεί συνέχεια, όπως και πέρσι. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω επιπρόσθετα στοιχεία. Θα ήθελα να αποφανθούν και οι συνάδελφοι έτσι ώστε το 2012 να υπάρχει ε, καλύτερη κατανομή των κονδυλίων μέσα στα πλαίσια των ε, 60 δις. Γιατί είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων, τις οποίες θα ορίσουμε επακριβώς εδώ. Ευχαριστούμε Λουίς Μακίνες και Μποναβία. Μακίνες πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και βεβαίως τον κύριο Καπούλα Σάντος. Του ευχόμαι και καλή επιτυχία στη δουλειά που έχει αναλάβει με τον προπολογισμό του 2012. Είναι, 12 είναι μια ε, δύσκολη προσπάθεια και σε σχέση με τον 2011, μέσα στο πλαίσιο αυτών των αντιπαραθέσεων και των διελκυστίνδων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ε, πιστεύω ότι τα καταφέρουμε καλά για τον προπολισμό του 2012. Σω είναι νωρί ακόμη να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα τα οποία γύρει εδώ ο Μάρκο είναι πολύ εύστοχα και πρέπει να μπουν στις προτεραιότητές μας. Ερωτώ λοιπόν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις ε, για το 2013 και τις άμεσες πληρωμές. Εάν υπάρχει κίνητρος δηλαδή για ε, εάν εξακολουθεί να επικρατεί ο κίνδυνος περί άρσης των αμέσων πληρωμών στα παλαιότερα κράτη-μέλη. Επίσης, το ζήτημα της ε, προσφοράς γάλακτος και φρούτων ε, στα σχολεία είναι πολύ, καινούριο, πολύ σοβαρό θέμα για μας, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Ε, τα καινοφανή τρόφιμα επίσης, δεδομένων και των τελευταίων προβλημάτων. Έχουμε επίσης τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής παράλληλα με αυτήν του προϋπολογισμού και έτσι χωρίς να είναι απαραίτητα συνδεδεμένα άμεσα τα θέματα ασφαλώς θα ανακύπτει το ένα στη συζήτηση του άλλου. Και ε, ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι πόσο η ασφάλεια των τροφίμων και τον, ε, και η γεωργική διάσταση είναι αλληλένδετες. Νομίζω ότι αυτά τα έχει αντιληφθεί ο κύριος Καπλός Άλτσος και θα τον ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λαβία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη συνάδελφο Μπαλτζάνη διότι μας παρουσίασε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη χρήση και γιατί θέλει να συμμετάσχουν όλες οι εξειδικευμένες επιτροπές εξ αρχής. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που συμμερίζομαι πλήρως, καθώς και η προσέγγισή της κατά την απαρχή του προϋπολογισμού με βάση τη στοχοθέτηση 2020. Ε, δηλαδή, ε, να δούμε πώς θα συσχετιστεί αυτή η στρατηγική με τους ετήσιους προϋπολογισμούς. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε και κάτι άλλο. Η πείρα μας πέρσι, με βάση τη δικασία προϋπολογισμού, μας ε, έδειξε και μας διδάσκει και κάτι νέο. Δηλαδή ότι από πλευράς ε, προϋπολογισμού μιλάμε για μείωση και αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών με βάση τον τομέα 2 υπαριθμών 2 του προϋπολογισμού. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε μεγάλο ενδιαφέρον και να προσέξουμε τη διαδικασία προϋπολογισμού με σωστές αξιολογήσεις. Δέχομαι την προσέγγιση της κυρίας Μπαλσάνη για προπαρασκευαστικές διαδικασίες για να δούμε ποιες είναι ποια είναι η καλύτερη ε, πύρα που αποκομίσαμε τα προηγούμενα έτη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι είναι δύσκολο ακόμα να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσει της αγοράς. Διότι όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά μόνο με το προσχέδιο προϋπολογισμού και το δεύτερο εξάμεινο με την αναθεώρηση της Κομισιόν θα έχουμε καλύτερη θεώρηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, θα ορίσουμε τις προτεραιότητες όπως είπαν οι Μαγκίνες, Σάντος και άλλοι. Και άλλοι και πολλές φορές υπάρχουν πολύ περιορισμένα περιθώρια. Όλοι μυρίσατε για το ε, πρόγραμμα φρούτα στα σχολεία, αλλά μιλάμε για 90 εκατομμύρια ευρώ και πέρα των 90 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούμε να κινηθούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλζάνη και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μία αποδοτική συζήτηση για τις προτεραιότητες. Ευχαριστούμε. Ε, Στεφάν Λεφόλ και μετά Ρέινερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Φραντσέσκα από την Επιτροπή Γεωργίας για να της πω ότι θα βρεθούμε στο πλευρό της για όλα όσα προτείνει για το 12 ως προς τον προϋπολογισμό που θα είναι αυτή τη φορά πολύ πιο μετρημένος και αυστηρός. Γιατί μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών θα έχει προβλήματα η Ευρώπη και πρέπει όλες οι επιτροπές να το καταλάβουν αυτό. Για μας είναι σαφές το πρόβλημα. Η γεωργία παραμένει τομέας και οικονομικός και δημιουργός θέσεων εργασίας αλλά Πρόκειται και για στρατηγικά θέματα, θέματα στρατηγικής, δηλαδή φαίνεται ότι αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίω δείχνουν ότι η τροφιμική ασφάλεια είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Η Φραντσέσκα ρώτησε τι προτεραιότητες πρέπει να έχει η Επιτροπή μας. Στη φάση αυτή βέβαια δεν έχουν προχωρήσει πολλοί συζητήσεις και Γι' αυτό θα περιοριστώ σε δύο-τρία θέματα. Ένα, η αγροτική πολιτική πρέπει να συμπεριλαμβάνει απολύτως τη στρατηγική 2020, ιδιαίτερα τα θέματα της, του περιβάλλοντος, της διατήρησης των πόρων και κάποιου επίπεδου ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. Για μας όμως η ΚΑΠ πρέπει να εγγράφεται τελείως μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Τώρα ιδιαίτερος η κτηνοτροφία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντική βαθιά κρίση και η κρίση αυτή μπορεί να κρατήσει πολύ. Το κόστος των ζωοτροφών αυξάνεται διότι αυξάνονται οι εντάσεις στις αγορές των δημητριακών και φοβάμαι ότι οι εντάσεις αυτές θα κρατήσουν πολύ καιρό και επομένως πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε και προτείνω σχετικά αντίθετα με αυτά που κάναμε για τον προπολογισμό του 11 αυτή τη φορά στον προπολογισμό του 12 δηλαδή να σκεφτούμε την περίπτωση ειδικών πόρων και ταμείων για την κτηνοτροφία. Όσο για τα πειραματικά ή πιλωτικά σχέδια Όλοι εδώ συμφωνούμε ότι πρέπει η Ένωση να κρατήσει τις δυνατότητες που έχει παρεμβάσεων στη Γεωργία. Ιδιαίτερα για το θέμα ενός ταμείου σταθεροποίησης που να επιτρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσει γρήγορα όταν σημειώνονται ή ξεσπούν σημαντικές κρίσεις στη Γεωργία. Να, Φραντσέσκα, Αυτά είναι τα τρία θέματα που ήθελα να σου γνωστοποιήσω μετά από αυτά που μας είπες σήμερα. Εντάξει Στέφανε, ο κύριος Ρέιμερς. Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την κυρία Μπαρτζάνη που ήρθε σήμερα να μας μιλήσει το Επιτροπή. Θα ήθελα να επισημάνω άλλη μια φορά ότι για τον προπολογισμό του 2012 όταν μιλούμε για θέσει εργασία στη Γεωργία θα πρέπει να ε, έχουμε πάντα υπόψη ότι δεν μιλάμε μόνο για τις γεωργικές εργασίες αλλά για μια σειρά από παράπλευρα επαγγέλματα και θέσει εργασία που εξαρτώνται από αυτήν και άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο μέγιστο να διαφυλάσσουμε αυτέ τι θέσει Για μένα πολύ σημαντικό είναι θέματα όπως και της μαθητείας ή της ε, κατάρτισης οι μετεκπαίδευση να μιλισμονηθούν επίσης γιατί μπορούν να επιτρέψουν κάποιον να ε, έχει περισσότερες ευκαιρίες να βρει ή να διατηρήσει τα εργασία του. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους φυσικά που θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούν ε, στη γεωργία στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να έχουμε την επόμενη γενναία που θα αναλάβει δραστηριότητα στην παραγωγή. Επίσης, Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε οικονομίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό δεν απαιτείται μόνο για τα πιο αδύναμα οικονομικά κράτη, αλλά για όλους. Και βεβαίως εμείς με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό έχουμε να δραματίσουμε και το ρόλο του παραδείγματος, του υποδείγματος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε να διαθέσουμε και ιδιαίτερα να συμφωνήσουμε στα κύρια θέματα, στους κεντρικούς άξονες οποίους θέλουμε να προαγάγουμε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ κύριο Τζορς Λάιον για τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Μπόλζα για την ε, παρέμβασή της. Θα ήθελα να ζητήσω διευκρινήσεις ε, για τα εξής. Την κυρία Μακίνες, μάλλον σχετικά με τα παρατηρήσεις της κυρίας Μακίνες, τις ε, οροφές, τα όρια δηλαδή για τις άμεσες πληρωμές και τι ε, προβλέπεται να γίνει εφέτος σε σχέση με τον... Ε, και βέβαια τι προβλέπεται και για το 2013 για... που είναι και το έτος για το οποίο εκφράζονται προς τις ανησυχίες. Επίσης, η κυρία Παλτζάνη μήπως θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για τα προγράμματα τα σχετικά με την ανάπτυξη πέθρου. Προχωρούν, υπάρχουν προβλήματα, Ξέρω ότι είναι βέβαια δύσκολο το θέμα δημοσιονομικά, είναι οι εποχές δύσκολες δημοσιονομικά, αλλά υπάρχει κάποια δυσκολία στην εκτέλεση, στην απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βαλτσάνη για τις απαντήσεις που μου δώσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για όλε αυτέ τι παρεμβάσει. Ο κύριο Αλτολόγκο να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Και στη συνέχεια ο Λούι και η Φρανσέσκα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ την κυρία Βαλτζάνη για την ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικά αιτήματα και ερωτήματα πώς ε, θα έχουν ε, οι άμεσες αναλήψεις πληρωμών για το 2012, δηλαδή κατά πόσο θα ισχύσει η δημοσιονομική πειθαρχία. Και το δεύτερο είναι τι, πώς θα έχει η εκτέλεση των πολιετών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Θα ήθελα όμως καταρχήν να πλαισιώσω τη συζήτηση. Δηλαδή αυτό το εγχείρημα προετοιμασίας του προϋπολογισμού 2012 που όπως ξέρετε θα εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στις 20 Απριλίου. 20-21 Απριλίου. Η διαδικασία προπαρασκευής και προετοιμασίας του προϋπολογισμού πλαισιώνεται από την οικονομική κρίση και τη μεγάλη πίεση των δημοσίων οικονομικών. Όμως θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμίσω, όπως ελέγχθηκε από άλλους ε, βουλευτές, ότι βρισκόμαστε στην ε, τελική φάση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 ε, και συνεπώς έχουμε χαμηλότερα περιθώρια ελιγμών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για την εκτέλεση των ε, πολιετών προγραμμάτων. και να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι προοπτικές για τον Γενικό Προϋπολογισμό του 2012. Φέτος προσδώσαμε μεγάλη προσοχή στις ε, δημοσιονομικές ανάγκες και παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην αγορά και τις προοπτικές ορισμένων γεωργικών αγορών μετά από τα διεθνή γεγονότα όπως της Βορείου Αφρικής και της Ιαπωνίας. Θέλουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο και τι επιπτώσεις υπάρχουν σε σχέση με τους κλειδονισμούς της αγοράς. Επίσης, είδαμε ποιες και πώς μπορούν να οριστούν οι οροφές σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές και το phasing in αυτών των επιδοτήσεων, ορισμένων δηλαδή επιδοτήσεων που θα ισχύσουν και για την επόμενη χρήση. Θα ήθελα λοιπόν να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής της δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν έχει λάβει αποφάσεις. Ετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό και εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή πριν από τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να ορίσει τις προτεραιότητες της. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτή την προθεσμία λοιπόν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τέτοιο νεφέλωμα στον ορίζοντα. Αλλά όπως είπαν ορισμένοι ευρωβουλευτές, το μέλλον είναι αρκετά δυσίων και ίσως χρειαστεί να εφαρμοστεί δημοσιονομική πειθαρχία. Ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε όμως. Ως προς το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, στο οποίο τη μεγάλη σημασία πολλοί βουλευτές. Θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό το θέμα και να πω τα εξή. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι με βάση το 2008, 2009 και 2010 οι πληρωμές ήταν χαμηλότερες από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στους αντίστοιχου προϋπολογισμούς για τις άμεσες πληρωμές. Πρέπει όμως να πω ότι επιτελέστηκε κάποια πρόοδος μετά το 2010 και έτσι έχουμε ελπίδες για το μέλλον. Δηλαδή, είδαμε αύξηση κατά 35% σε σχέση με το 2009 ως προς το ρυθμό εκτέλεσης. Για την περίοδο 2007-10, το σύνολο των πληρωμών, δυνάμει αυτών των προγραμμάτων, είναι της τάξης των 38 δις ευρώ δηλαδή 39,5% του συνόλου του δημοσιονομικού πακέτου για την περίοδο 2007-2013. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι εκτιμήσεις από τα κράτη-μέλη για το 2011 μας οδηγούν στο 13,7 σε 13,7 δις που πρέπει να συγκρίνουμε με τα 12,2 δις, τα οποία προβλέπονταν αρχικά στον προϋπολογισμό. Και αυτό αφορά και τις μεταφορές. Άρα, δεν θα υπάρχει ε, μειωμένη χρήση για το 2011. Άρα υπάρχουν θετικές πρόπτικες που μας επιτρέπουν να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων mm. και εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των κρατών μελών, τότε το 2011 και 2012 θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας απάντησα εμπεριστατωμένα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε. Άλτο, δεν ξέρω ε, κατά πώς απαντήσατε πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ε, δυσίωνες οι προοπτικές. Ε, ο Λουίς πρώτα και η Φρανσέσκα μετά. Ο Λουίς πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, απλώς θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να σταθούμε στις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις και θα πρέπει να γίνει μία σωστή εκτίμηση σε σχέση με τις αρχικές μας προτάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει θετική ή αρνητική αποτίμηση των ε, πρωτοβολιών μας και κατά πόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ε, γίνεται σωστή ένταξη των προτεραιοτήτων μας. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με τα συνολικά ποσά που προτείνονται. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με την εκτέλεση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για να δούμε κατά πόσο αυτός ο χαμηλός ρυθμός εκτέλεσης έχει να κάνει με την χρηματοοικονομική κρίση. Δηλαδή, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα, δημοσιονομικά προβλήματα και έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να απορροφήσουν τα κοινοτικά κονδύλια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ε, συνολική μας σχέση, ε, σκέψη και συλλογιστική ως προς την συγχρηματοδότηση. Και αυτό αφορά την ε, χρηματοοικονομική κατάσταση σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπαλτσάνη, τους συναδέλφους και θα ορίσουμε και τη δική μας στρατηγική για να προβάλλουμε μία καλώς διαρθρωμένη πολιτική για το επόμενο έτος. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Λουίς ή Φραντσέσκα, για τα συμπεράσματά της. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος Καπούλα Σάντος σε σχέση με την προπαρασκευαστική δάση και τα πλειοτικά σχέδια. Χρειάζεται μια προσεκτική ανάλυση αυτού του πακέτου για να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούμε τα ευέλικτα περιθώρια που υφίστανται και για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Εάν λάβουμε υπόψη την αξιολόγηση της ε, Κομισιόν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι θετική για πολλά πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Άρα θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν πριν από το καλοκαίρι να υποβάλουμε έναν κατάλογο για τα σχέδια και τις δράσεις και θα είναι ο, πιο, ο πρώτος τομέας παρέμβασης σε σχέση με τις προτεραιότητες και τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής. Άκουσα με προσοχή όλες τις παρεμβάσεις και νομίζω ότι, ότι η ε, Λεφόλ και ο Στέφανο Λεβία μας ε, τόνισαν την διάσταση της γεωργίας που θα κινηθεί προς μια νέα κατεύθυνση. Διότι ανακύπτει όχι το θέμα της εργασίας, αλλά και της στρατηγικής του 2020, δηλαδή η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο για να έχουμε σημεία επαφής, ήδη επαφής, τα οποία να είναι πραγματικά καινοτόμα. Ευχαριστούμε τη Φραντσέσκα. Άρα έχει λήξει και το 12. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά, διότι περιμένουμε τον Ντάτσαν Τσόλο, τον Επίτροπο, ο οποίος θα προσέλθει εδώ για μία ανταλλαγή απόψεων. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Riprendiamo. Να καλωσορίσουμε τον ε, Επίτροπο Ντάτσον Τσόλος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας για το 2012. Βεβαίως το 2012 θα επικεντρωθούμε στην ε, αναθεώρηση της ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος θα μας υποβάλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και άλλα σημαντικά σχέδια για τη γεωργία το 2012. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ακούσουμε τον Επίτροπο ο οποίος είναι μαζί μας σε αυτή την Επιτροπή και θα προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για το χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Ντάτσαν έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να συζητήσουμε ήδη από τώρα τις προτεραιότητες για το 12. Η Κομισιόν ως συνήθως θα ετοιμάζει το πρόγραμμά και θα το υποβάλει εγκαίρως, αλλά ήδη από τώρα μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα κυριότερα στοιχεία της. Ιδιαίτερα όλα όσα διαπιστώσαμε πέρυσι. Καταρχήν θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη έχει υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας στα πλαίσια των προβλεπομένων από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από την πρώτη ανάγνωση ορισμένων νομοθετικών προτάσεων φάνηκε ότι η διαδικασία της συναπόφασης ε, λειτουργεί πολύ καλά. Παραδείγματο χάρη οι δέσμοι για το εμπόριο της βανάνης και των υνοπνευματοδών. Ε, Όπως είπε και ο Πάολο, το κυριότερο στοιχείο που μας απασχολεί αυτή τη φορά είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Η έκθεση ΛΑΙΟΝ ακολουθήθηκε από τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν και τώρα προετοιμάζουμε την νομοθετική δέσμη. Ξέρω ότι και εσείς συζητάτε τα θέματα αυτά έντονα, την έκθεση DES ας πούμε. Το Συμβούλιο επίσης προετοιμάζει τα συμπεράσματά του. Οι νομοθετικές προτάσεις που θα ακολουθήσουν για την ΚΑΠ του 13 θα υποβληθούν στο δεύτερο ήμιση του έτους, το φθινόπωρο, μετά από την παρουσίαση των δημοσιονομικών προοπτικών, των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών που θα γίνει τέλη Ιουνίου. Η νομοθετική πρόταση για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη αυτή μετά τις δημοσιονομικές προοπτικές μαζί με άλλα σημαντικά θέματα που θα υποβάλει η Κομισιόν όπως είπα τον, το φθινόπωρο, για να προλάβει εντωμεταξύ την αξιολόγηση που ετοιμάζει επίσης τον Ιούνιο. Πρέπει επίσης να τονίσω ποια, νομοθετικά, ποια νομοθετήματα προετοιμάζονται, ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας ιδιαίτερα οι δέσμοι για την ποιότητα και οι δέσμοι για τα γαλακοτοκομικά. Και εδώ η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την έγκριση από την πρώτη ήδη ανάγνωση ή δυνατόν. Και Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι και η δική σας συμβολή Νίκολσον για τα γαλακτοκομικά, Γκαρθία Περές για την ποιότητα. Για το 2012 λοιπόν θα γίνει η συζήτηση για τις νομοθετικές προτάσεις, όλες αυτές τη δέσμη, που θα μας απασχολήσει μέχρι τα τέλη του 12. Οι προτάσεις θα γίνουν το ξαναλέω το φθινόπορο και μετά θα αρχίσει η κυρία συζήτηση. Πέρα από αυτό όμως, όπως είπα και κατά τις ακροάσεις μου, θα έρθω να σας δω και ως προς μια νέα πρωτοβουλία γιατί φέτος θέλω να γίνει δημόσια διαβούλευση για την πολιτική προώθηση των γεωργικών προϊόντων διότι θεωρώ ότι η προώθησή τους πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη και καλύτερα δομημένη στα πλαίσια της κάποια για διάφορους λόγους. Πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες του ανοίγματο ορισμένων αγορών και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται διεθνώς η υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, στην ποιότητα των τροφίμων μας. και αυτό να προωθηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα διεθνώς. Ταυτόχρονα όμως να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και στην ευρωπαϊκή αγορά, στην εσωτερική αγορά. Ζήτησα λοιπόν από τις υπηρεσίες μου να κάνουν, να υποβάλουν προτάσεις επί τη βάση αυτών των ιδεών και πριν το καλοκαίρι προτείνω να δημοσιευτεί μια πράσινη βίβλος για την προώθηση αυτή των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και μετά στις αρχές του επόμενου έτους να κάνουμε μια ανακοίνωση με τα συμπεράσματα αυτής της διαβούλευσης ή πρασίνης βίβλου ώστε να προκύψουν από αυτήν συμπεράσματα, προτάσεις και για τον προϋπολογισμό και το 12 επίσης πριν λήξει το 12 να κάνουμε μία νομοθετική πρόταση που να καθορίζει το γενικότερο νομοθετικό νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να οικοδομηθεί αυτή η πολιτική προώθησης στα πλαίσια της ΚΑΠ. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη απάντηση, ανταπόκριση σε όλα όσα έχουμε πει και ακούσει για τα προβλήματα του αγροτροφημικού τομέα και της έμφασης που θέλουμε να δώσουμε στην ποιότητα των προϊόντων και στην δημιουργία νέων δικτύων διανομής πιο αποτελεσματικών. Γι' αυτό χρειάζεται το κατάλληλο νομοθετικό νομικό πλαίσιο. Επίσης με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι οι δασμοί μειώνονται για ορισμένα τρόφιμα και αν θέλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεργαστεί με τα σχέδια που ανέφερα, με τα χαρά θα δεχτούμε. Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία που μπορώ να σας προτείνω. Καταλήγω ότι το 12 θα ήθελα να σκεφτούμε το θέμα αυτό της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ νομοθετικά με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα αυτή πρόταση της προώθησης των ευρωπαϊκών αγροτροφημικών προϊόντων. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ντάτσαν. Πλούσιο το πρόγραμμα που μας παρουσιάζεις και ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Έχουμε μέχρι τις 12.30. Μέχρι τις 12 μάλλον. Περιθώριο όπου θα πρέπει μετά να αποχωρήσει ο κύριος Επίτροπος. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι. Έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους. Ο κύριος Δέσ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που, έκανε την, ε, που ήρθε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας για να μας ενημερώσει για τη δουλειά του και να συζητήσει τα θέματα αυτά μαζί μας. Ως ηγητής για τις νέες κατευθύνσεις γεωργικής πολιτικής έχω καταθέσει την έκθεσή μου, την οποία μπορούμε και να συζητήσουμε τώρα, δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε την κατεύθυνση προς την οποία μπορούμε να προχωρήσουμε και προκειμένου να βελτιώσουμε τις ε, ε, προτάσεις αυτές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο στόχος της, ε, της χάραξης μιας πολιτικής με προοπτική το 2013. Είναι ένας στόχος κοινό πιστεύω, ένας στόχος τον οποίο επιδιώκουμε όλοι από κοινού και η κοινή γεωργική πολιτική από το 2013 πρέπει να διασφαλιστεί, ε, να διαφυλαχθεί και θέλουμε ταυτόχρονα χάρη στην γεωργία στην Ευρώπη να εξασφαλίσουμε και βιώσιμη καλλιέργεια, βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων μας. Υπάρχουν βέβαια διαφωνίε ω προ κάποια τεχνικά θέματα όπω το screening για το θα πρέπει να επαχθεί στον πρώτο η στο δεύτερο πυλώνα. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτό θα εκριθεί η μάχη. Στόχο μα και πρωταρχική προτεραιότητα, και το βλέπω αυτό και στι συνομιλίε με του γεωργού, είναι να αποφύγουμε την γραφειοκρατία και του να καταστήσουμε πιο απλό το σύστημα. Εγώ πολύ ευχαριστώ θα ακούσω όποια πρόταση έχει σαν στόχο ακριβώ αυτό το θέμα, την απλούστευση δηλαδή, ε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα προστευμένο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο θα ικανοποιεί του στόχου που από κοινού έχουμε προσδιορίσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ καλή συνεργασία την οποία μα έχετε προσφέρει και καλλιεργείτε πάντοτε εδώ και χθες ε, κύριο Σμπαρόντε Κάστρο ο πρόεδρος μας ε, μας μίλησε για τις προσπάθειες τις σχετικές με την πρόοδο στην εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων της Συνθήκης Λισαβόνας έτσι ώστε ε, να έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας ορθολογικό και αποτελεσματικό. Περιμένω να ακούσω τις απόψει των συναδέλφων ε, στα θέματα της δικής μου πρότασης. Είμαι πάντα πολύ φιλομαθής και ε, περιμένω να ακούσω τι έχουν να μου πούνε οι συνάδελφοι για να επηρεαστώ από τις απόψεις τους πιστεύω ότι μπορούμε έτσι να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή πρόταση για τις προσεχείς ε, για τις προσεχείς διαστάσεις ε, και πτυχές της γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριο Σκαπουλασάντος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή μας. Όπως είπατε πολύ σωστά, ε, θα έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη αναθεώρηση με μια μεγάλη αναθεώρηση της πολιτικής της ΚΑΠ και όπως είπαν οι σοσιαλιστές θα πρέπει να φτάσουμε σε μια ευρεία ε, συνένεση έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα λειτουργικά πλαίσια μέσα στα πλαίσια της συναπόφασης για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τις ε, απόψεις μας, αλλά ένα συμβιβασμός σημαίνει ότι δεν θα μας επιβληθούν οι απόψεις των άλλων αποκλειστικώς. Η σοσιαλιστική ομάδα ασχολήθηκε εις βάθος με το θέμα. Υπάρχει μεγάλη εσωτερική συνοχή. Ήδη έχουμε φτάσει σε έναν προσυμβιβασμό ως προς τα θέματα που μας απασχολούν για να μειώσουμε τον αριθμό των τροπολογιών και για να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά ζητήματα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια δυνατή ΚΑΠ και να έχουμε και μια διαπραγματευτική θέση η οποία να είναι αποφασιστικής ε, σημασίας. Προσδοκούμε αυτό το καλό αποτέλεσμα και ελπίζουμε ότι το νομοθετικό κείμενο θα εντάξει και τα δικά μας θέματα ως προς τα άλλα θέματα, δηλαδή το ποιοτικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό και θα ασχοληθούμε και με αυτό και βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε και τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε κύριε Επίτροπε σε σχέση με την ε, πρωτοβουλία για την πρόθεση αγορατικών προϊόντων. Έτσι θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε για να δώσουμε μία συνέχεια σε αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Τέλος, θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στον ε, κύριο Επίτροπο είπαμε ότι θα αρχίσουμε τη συζήτηση για το προϋπολογισμό του 2012 και τώρα θα ορίσουμε τις δικές μας προτεραιότητες επειδή δεν έχουμε ακόμα μία πρόταση από την Εκτελεστική Επιτροπή, θα εκτιμήσουμε την κατάσταση ανάλογα με τα πολιτικά προσδοκόμενα και θα λάβουμε υπόψη βεβαίως και τα διεθνή γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις αγροτικές τιμές, όπως η κατάσταση στη Βόρειο Αφρική και το, ε, με την τραγική κατάσταση και τα μεγάλα, τα μεγάλα ατυχήματα στην Ιαπωνία. Περιμένουμε λοιπόν μία ε, αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετά θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο οι προοπτικές του 2012 μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση και κατά πόσο η Επιτροπή διαθέτει ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην χαρακτηριοποίηση αυτής της κατάστασης και στον προσδιορισμό της για να ορίσουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Ευχαριστώ. Ο George Lyon. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλωσορίζω τον Επίτροπο Τσόλος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Με χαρά σας βλέπουμε εδώ. και εσάς και την παρουσίαση για το έτος 2012. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πράγματι θετικό αποτέλεσμα σε, στον τομέα εκείνων των καρόνων της ε, Συνθήκης Λισαβόνας που υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ ιδιαίτερα εκτιμώ αυτή την ε, πρόοδο που σημειώνεται. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταθέσω κάποιες ερωτήσεις προς εσάς που έχουν να κάνουν με τα θέματα ε, της εισαγωγικής σας παρέμβασης ως προς τις νομοθετικές προτάσεις που λέτε πως προβλέπετε να καταθέσετε το φθινόπωρο. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Φθινόπορο σημαίνει Αύγουστο-Σεπτέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεστε για αυτές τις προτάσεις. Και δεύτερον, Στι μεσονομικέ προτάσει τη Επιτροπή για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρόκειται για ένα λεπτομερές έγγραφο. Θα καταθέσετε δηλαδή συγκεκριμένα ποσά για κάθε μία από τις θέσεις του προϋπολογισμού. Ή θα ορίσετε μόνο προτεραιότητες. Γιατί έχει διαρρεύσει ένα σχέδιο εγγράφου πριν από 18 περίπου μήνες, το οποίο έδειχνε πως ε, πρόκειται να κατεθούν μάλλον προτάσεις προτεραιοτήτων και όχι συγκεκριμένες προτάσεις Επιτροπής για δαπάνε σε κάθε θέση του προϋπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το έγγραφο των δημοσίευτων τον Ιούνιο. Οι προτάσεις για προαγωγή των γεωρικών προϊόντων με νέα ποσά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσε και θα θέλαμε πιο συγκεκριμένε προτάσει να ακούσουμε για τα ευρωπαϊκά βέβαια προϊόντα και την προαγωγή του και σε, η προβολή του και σε άλλε αγορέ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα θέλαμε να δούμε συγκεκριμένα τι εννοείται, αλλά βέβαια μα ενδιαφέρει και η εμπορευματοποίηση ή η προώθηση καλύτερα των προϊόντων μα και μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά καλύτερα. Άλλο ένα θέμα, το οποίο δεν θέξατε εσεί, αλλά το κρίνω πολύ σημαντικό, και το λέω μια και είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Επίτροπο Ντεγκιούχτ πριν από δύο εβδομάδε περίπου, ο οποίο μου εξήγησε πω η Επιτροπή ελπίζει να μπορέσει να υποβάλει πρόταση προσφορά προς τις χώρες Μερκοσούρ για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Μάλιστα μου είπε ο κύριος Νταγκίχτ ότι ε, το δικό σας ε, επιτελείο, εσείς προσωπικώς έχετε την ευθύνη για την συζήτηση της δυνατότητας πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις χώρες Μερκοσούρ στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και του Τούμπαλιν. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, έχει ολοκληρωθεί το σχετικό έργο, έχετε δηλαδή ολοκληρώσει τους όρους με τους οποίους θα αποβληθεί αυτή η προσφορά και έχετε μελετήσει τι είδους συνέπειες θα έχει στην αγορά των κρατών αυτών και, τον, και τη δική μας βέβαια ε, αυτή ε, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών για τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, τουλάχιστον για τη Σκοτία, αλλά φαντάζομαι ότι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έχετε συζητήσει, έχετε μελετήσει τι συνέπειε στη δική μας παραγωγή, τη παραγωγή η οποία δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στη μεγάλη πίεση των φθηνών εισαγωγών από τη Βραζιλία και την Αργεντινή κυρίω. Έχετε κάποιο αντιστάθμισμα ή μπορείτε να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμφωνία αυτή με τις χώρες Μερκοσούρ, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ, όπως και οι άλλοι συντονιστές, ε, τον κύριο Τσόλος. Με χαρά σας βλέπουμε και πάλι εδώ. Με χαρά ακούμε τις προτάσεις σας για τις προτεραιότητες του μέλλοντος. Πολλά είναι τα θέματα νομίζω πρέπει να καλυφθούν. Πολλά είναι τα θέματα στα οποία βλέπουμε ή περιμένουμε να δούμε τις δικές σας προτάσεις για τη μεταρρύθμιση. που είχε προταθεί αρχικά για Ιούνιο-Ιούλιο και τώρα μετακυλείεται προς το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί άλλη μια αναβολή, θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί όσο βέβαια καθυστερεί η υποβολή τη πρόταση, τόσο πιο δύσκολο είναι για μα και πιο στενά τα περιθώρια για να συμμετάσχουμε, να συμβάλλουμε σε αυτήν με τι δικέ μα προτάσει. Επίση, Θεωρώ ευπρόσδεκτο το γεγονό ότι θέλετε να βοηθήσετε στην προαγωγή των ευρωπαϊκών προϊόντων. Πιστεύω ότι αυτό είναι διτό εγχείρημα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβάλλουμε τα προϊόντα μα, αλλά και έξω από αυτήν. Και θα ήθελα να δω κάποιε καινούριε ιδέε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλέ οργανώσει και φορεί οι οποίοι θεσπίζονται για την προβολή των προϊόντων, τουλάχιστον στη δική μου πατρίδα, και έχω πολλέ αμφιβολίε για το κατά πόσον δαπανώνται φρόνημα τα χρήματα αυτά, τουλάχιστον από ορισμένου που δραστηριοποιούνται σε αυτού του φορεί. Έτσι λοιπόν πιστεύω πρέπει να επανεξεταθιστεί αυτή η υπόθεση. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ε, και χώρος για την προβολή. Ε, μια γεωργική έκθεση, φερειπίνη, έκθεση γεωργικών προϊόντων αρκεί, και που ο καθένας έχει το δικό του περίπτερο και βάζει τα προϊόντα της ε, περιοχής του, της περιφερεια του, της περιφερειάς του. αρκούν όλα αυτά ή πρέπει να κάνουμε κάποια διαφορετική επιλογή. Και επίση περιμένουμε να δούμε και να συζητήσουμε όλοι μαζί το πακέτο των μεταρρυθμίσεων για να έχουμε την ευκαιρία, όπω είπα και το Κοινοβούλιο, με την έκθεσή του να ε, κάνει τι προτάσει του. Ο κύριος Πεκαπλού Σάντους επισήμανε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις από πλευρά των μελών της Επιτροπής μας για το τι μορφή θα πρέπει να λάβει αυτή η μεταρρύθμιση και προς τα που πρέπει να κινηθεί. Αυτό είναι θα έλεγα μια μετριοπαθή ε, παρουσίαση της κατάστασης. Εν πάση περιπτώσει όμως νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα τι θέλει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα το κύριο αίτημα είναι η απλούστευση απλούστευση στη γραφειοκρατία, στη διοίκηση, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που διεκδικεί ο πολίτης και κυρίως ο γεωργός ε, στην Ευρώπη. Ωστόσο, εγώ βλέπω και κάτι άλλο. Ότι κάθε φορά που γίνεται μια μεταρρύθμιση δεν διαγράφονται αντίστοιχες πτυχές της προηγούμενης ρύθμισης οι οποίες επιβάλλουν υπερβολικό φόρτο και δεσμεύουν πολύ στην ε, ε, δράση του τον παραγωγό, τον γεωργό ή τον κτηνοτρόφο. Σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση λοιπόν. Και επίση μην γελιόμαστε. Ο αγώνα θα κρυθεί πάνω στην παράγραφο 22 τη έκθεση ΔΕΣ και στο πρασίνισμα του τέταρτου πυλώνα. Εγώ θα επισημάνω ότι δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πιο πολύ πρασίνισμα ο τέταρτο πυλώνα. Πρασίνισμα χρειάζεται ο δεύτερο πυλώνα. Αν είναι να δώσουμε πιο πολύ οικολογική διάσταση, στο δεύτερο πυλώνα λοιπόν, κύριε Τσόλο. Εκεί θα πρέπει να δώσετε την έφαση. Και θα σα πω και κάτι άλλο κύριε Πέτροπα. Ότι καλό θα ήταν η Επιτροπή, κατά την άποψή μου, να είναι πιο ανοιχτή εναντί του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι παραμένετε κρυψίνοε εναντί Μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ ε, ο καθένας από την περιφερειά του, από το χωριό του, από την περιοχή του, με τις προτεραιότητες του και τις γνώσεις του. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε ή να παρεμποδίσουμε την έρευνα, την ανάπτυξη, τις προτάσεις οι οποίες απαιτούνται, απαιτείται να κατατεθούν και να αναπτυχθούν προκειμένου να ε, έχουμε μια καλή γεωρική πολιτική μετά το 2014. Καθόμαστε εδώ και συζητούμε για την ασφάλεια των τροφίμων, της προμήθειας των τρόφιμων. Και μπορεί να έχω καταλήξει λάθος ε, συμπέρασμα και διορθώστε με, μακάρι να με διορθώσετε δηλαδή. Αλλά φοβούμαι ότι σε 12 μήνε θα ξαναβρεθούμε στην ίδια αίθουσα να συζητούμε ακόμη μεγαλύτερου κινδύνου για την ασφάλεια τη ε, προμήθεια σε τρόφιμα, ε, με ακόμη δυσμενέστερε συνθήκε. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε όλοι να διαδραματίσουμε ένα ρόλο επικοδομητικό. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, Εθνικά Κοινοβούλια και Εθνικέ Κυβερνήσει. Όλοι βέβαια λένε ωραία λόγια και μεγάλα λόγια για την ε, προμήθεια στα τρόφιμα και την ασφάλεια αυτή, αλλά στην πράξη δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Όταν ήρθα εγώ το 91 στο Κοινοβούλιο σε ευρωβουλευτή και πρόεδρε τελειώνω εδώ, είχαμε ε, λίμνες γάλακτος, βουνά κρέατος και λόφου βουτύρου. Τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τουναντίον αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα σπάνιδας τροφίμων και αυτό ακριβώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λοράνσο Φοντάνα. Sorry, Martin Oschling first, and then Fontana. Πρώτα Όσλινγκ. Χόισλινγκ. Κακό δείγμα να παραβλέπετε τους πρασίνους στη σειρά των ομιλητών, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι να σας βλέπω εδώ. Όντω νομίζω ότι η παρουσίαση εδώ και η συζήτηση που γίνεται μπορεί να βοηθήσει στην ε, περαιτέρω προαγωγή ακόμη του διαλόγου. Βεβαίω θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν καλύτερη προβολή των ευρωπαϊκών ε, γεωργικών προϊόντων με ένα μήνυμα διαφημιστικό ε, ώστε να εξηγούμε λίγο πολύ στον καταναλωτή τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το δικό μα ευρωπαϊκό προϊόν από το εισαγόμενο γεωργικό προϊόν. Και ακριβώ εδώ έχουμε να κάνουμε και με, τους, με τη βασική μας στόχευση στην μεταρρύθμιση γεωργικής πολιτικής. Τις προδιαγραφές, τις οποίες δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει και οι οποίε αποτελούν στη τελευταία ανάλυση το κύριο χαρακτηριστικό, το σημάδι που χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά και γεωργικά προϊόντα. Εδώ λοιπόν στη γεωργική ε, πολιτική στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ε, παρά τις πιέσεις για εκβιομηχάνηση και εντατικοποίηση, κυρίως στην κτηνοτροφία που ασκούνται με ιδιαίτερη ένταση τον τελευταίο καιρό. Έχουμε τη συζήτηση στη Γερμανία βεβαίως, αλλά αναπτύσσεται και η αντίστροφη τάση για το τι μπορεί να συμβεί στη Γεωργία και το τι τελικά επιδιώκουμε από τη γεωργική μας παραγωγή. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος ε, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει για τη γεωργική μεταρρύθμιση στόχους σαφείς, στόχους που κρίνω θετικούς Ήδη το Νοέμβριο σημειώθηκε συνένεση πάνω στο πρόγραμμα, στην προ... στις προτάσεις σας, στο έγγραφό σας και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Επίσης, υπάρχει μια πρωτοβουλία, πιστεύω, για το cupping παρά τις ε, πιέσεις ε, των κρατών μελών που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη δημοσιονομική πολιτική και πρέπει από αυτή την έννοια να αντιμετωπιστεί, να, να, να προβληθεί το θέμα αυτό, γιατί καλό θα είναι να μην παραβλέπουμε τις πραγματικότητες και τις δημοσιονομικές να συστούμε για τη γεωργική πολιτική. Μερικές φορές έχουμε την τάση τη γεωργική πολιτική να κάνουμε προτάσεις οι οποίες ξεπερνούν τις δυνατότητες μας ε, τις ε, δημοσιονομικές Και βέβαια ξέρουμε ότι η Γεωργία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επί του προπολογισμού, απορροφά μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού μα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συζητηθούν και βέβαια μέσα στι πολιτικέ μα ομάδε. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο Άλμπερτ Πάντοτε είναι πρόθυμο για συμβασμό, πράγμα το οποίο χαιρετίζω. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις πολυάριθμες τροπολογίες, οι οποίες πάντα δεν βοηθούν στο να καταστεί πιο σαφές το κείμενο. Ε, ενώ εμείς θέλουμε ένα κείμενο το οποίο θα τα γράφει ξεκάθαρα τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό καλό θα είναι να μην παρασυρθούμε σε πολλές ε, τροπολογίες οι οποίες τελικά θα ε, μας κάνουν να χάσουμε το στόχο της συζήτησης. Χτες έγινε μια συζήτηση και για τα μέτρα στην αγορά, για τους κανόνες. Συζήτηση που θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. Γι' αυτό απευθύνω για άλλη μια φορά έκθεση, έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει καινούριες προτάσεις για τα μέτρα τα σχετικά με τη λειτουργία των αγορών. Υπάρχει και το θέμα βέβαια τη ασφάλιση που συζητήσαμε πάλι και χθε, αλλά δεν μπορούμε να το λησμονούμε. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ούτε την οργάνωση και τα μέτρα τα σχετικά με την οργάνωση των αγορών, ούτε την ασφάλιση όπως και στην περίπτωση του γάλακτος συγκεκριμένα, έχουμε να κάνουμε με την διαφύλαξη του εισοδήματος πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γαλακτοκομικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ε, υπάρχει κίνδυνος με την ε, προόδο της απελευθέρωσης να κινδυνεύσουν πολλές από αυτές τις ε, επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα. Επίσης ακούστηκε νωρίτερα ε, το ζήτημα από τον κύριο Νίκολσον, το ζήτημα της ασφάλειας στην ε, προμήθεια τροφίμων και γενικά το ζήτημα το επιστηστικό παγκοσμίω σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και έτσι και στις εισαγωγές τροφίμων, από τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε να απαλλαγούμε, από τις οποίες εξαρτώμεθα ακόμη, ε, τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στην προμήθεια τροφίμων που θα πρέπει να συζητήσουμε, το οποίο θα πρέπει να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αποκόψουμε και από τον προβληματισμό το σχετικό με τη γενετική ε, μηχανική, με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δηλαδή, και γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει και στην ε, μεταρρύθμιση της ιωρικής πολιτικής να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Περιμένω εδώ τις απαντήσεις του ε, Επιτρόπου. Ναι, βεβαίως. Ε, σήμερα μας απασχολεί η ατζέντα σχετικά με το 2012. Δεν θα ήθελα να επιβαρύνουμε τη συζήτηση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Λορέντσο Φοντάνα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι παρόν εδώ και συμφωνώ όταν μιλά για την προώθηση των προϊόντων μας ιδιαίτερα σε σχέση με την ευρωπαϊκή παραγωγή, σε σχέση με το υπόλοιπο του πλανήτη. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με αυτά που είπε ο George Lyon. δηλαδή τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και υπολείπου κόσμου, ιδιαίτερα στις σχέσεις μας με το Μερκοσούρ. Γιατί πάντα Δυστυχώς τα προϊόντα που εισάγουμε από τρίτες χώρες δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με την ποιότητα των δικών μας προϊόντων και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωργική μας παραγωγή. Άρα, αυτό το κριτήριο υφίσταται εν υπάρχει και στις προτάσεις για την ΚΑΠ. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου η Ευρώπη να επιβάλλει στα εισαγόμενα προϊόντα να έχουν τις ίδιες ποιοτικές ε, παραμέτρους. Ευχαριστούμε πολύ Λορέντσο γιατί ε, παρέμεινες και σε λογικά χρονικά πλαίσια. Ρουμπίχα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριο Ρούμπιξ. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ήρθατε να μας επισκεφθείτε στην Επιτροπή μας, να μας μιλήσετε. Βλέπουμε ότι είστε πάντοτε διαθέσιμος για συνεργασία και ε, συνομιλία μαζί μας και διάλογο. Απλώς θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μετατραπεί αυτός ο διάλογος σε μια απλή επανάληψη, γιατί βλέπουμε τα θέματα να επανέρχονται διαρκώς. Επί παραδείγματι ε, το ζήτημα των άμεσων πληρωμών. Είναι ένα ζήτημα που έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαίο πολίτη, για το δικό μου τουλάχιστον ψηφοφόρο και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εάν ε, στο μελλοντικό πρόγραμμα της ε, Επιτροπής έχετε υπόψη να ε, μιλήσετε για τις άμεσες πληρωμές και την εξίσωση των άμεσων πληρωμών στους παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Επίτροπος παρακαλώ να λάβει το λόγο για να δώσει απαντήσεις και μετά θα επανέλθουμε. Παρακαλώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ε, χρονοδιάγραμμά μας, με, την μας, με το πρόγραμμά μας, κυρίως με τη μεταρρύθμιση Κυρίω με τη μεταρρύθμιση, λοιπόν, ξέρω ότι έχω να δώσω κάποιε απαντήσει, αλλά τι συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσει θα δείτε με την υποβολή τη νομοθετική πρόταση. Πότε θα κατατεθεί η νομοθετική πρόταση συγκεκριμένα. Είπα φθινόπωρο, γιατί είμαστε τώρα στη φάση τη επεξεργασία νομοθετική πρόταση. Έχουμε ξεκινήσει με τι μελέτε επιπτώσεων των διαφόρων στοιχείων περιλαμβάνει, που θα περιλαμβάνει αυτή η ε, πρόταση, νομοθετική πρόταση. Ωστόσο θα αντιλαμβάνεστε κι εσεί ότι πρέπει να έχουμε και τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, τουλάχιστον κάποιου προσανατολισμού των δημοσιονομικών προοπτικών για να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η νομοθετική πρόταση. Ε, άπαξ και, δημοσιοποιηθούν, δημοσιευθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές, πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε αυτές τις μελέτες επιπτώσεων για να έχουμε και την επιχειρηματολογία μας υπέρ της μίας ή της άλλης λύσης που θα προτείνουμε με την ε, ε, νομοθετική πρόταση. Η μελέτη επιπτώσεων ασφαλώς απαιτεί κάποιο χρόνο. Έτσι λοιπόν, εάν μέχρι τα τέλη Ιουνίου-Ιουλίου έχουμε τις λύσεις, τις ε, απαντήσεις για τη μελέτη επιπτώσεων και υπενθυμίζοντα ότι ο Αύγουστο είναι ούτω ή άλλω διακοπέ, χαμένο χρόνο λίγο πολύ. Μετά έχουμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να τελειοποιήσουμε, για να ολοκληρώσουμε τι νομοθετικέ προτάσει και να δούμε μέσα από τη διαβούλευση με τι ε, ε, υπόλοιπε υπηρεσίε πώ βλέπουν εκείνε, κάθε μία χωριστά, τι επιπτώσει του προπολογισμού του αυτή τη νομοθετική πρόταση. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να προσανατολιζόμαστε μάλλον προ τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, λαμβανωμένη υπόψη τη περίοδου των θερινών διακοπών και τη ανάγκη για διαβούλευση μεταξύ των διαφορών τμήματων και υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μέχρι τώρα και πάλι βάσει των προτάσεων του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι, δηλαδή δημοσιονομικές προοπτικές να έχουν κατευθυνθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή αρχά Ιουλίου με αυτό το δεδομένο. Τη λεπτομέρεια των ε, δημοσιονομικών προοπτικών δεν μπορώ φυσικά να την ε, εκθέσω εγώ. Ο κύριο Λεβαντόφσκι που είναι ο αρμόδιο τη γνωρίζει καλύτερα από όλου και μπορεί να δώσει απαντήσει. Ξέρω ότι θα την παρουσιάσει στο συλλογικό όργανο τη Επιτροπή ω προ το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων ε, που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή. Πιο πολλέ λεπτομέρειε δεν μπορώ να δώσω. Πάντως, φαντάζομαι ότι μπορώ να ε, αντλήσω όταν είναι έτοιμος ο κύριος Λεβαντόφσκι τις, ε, το πλαίσιο στο οποίο μπορώ εγώ να προχωρήσω στι δικέ μου προτάσει. Αλλά όπω είπα, δεν μπορώ τώρα να σα δώσω συγκεκριμένε απαντήσει, γιατί είναι αρμοδιότητα του κύριου Λεβαντόφσκι ο οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των δημοσιονομικών προοπτικών. Ακόμη δεν έχει συζητηθεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή συλλογικού Συλλογικό Όργανο. το σχέδιο περί προβολής των ευρωπαϊκών προϊόντων. Πάλι δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα. Ίσως αντελήφθητε κι εσείς ότι η στόχευσή μου είναι σε κάθε κύκλο ε, διαβούλευσης και παρουσίασης της ε, προτάσεως να ε, γίνει ο διάλογος των δυνατών πιο ανοιχτό. Με μια πράσινη βίβλο θα ξεκινήσουμε για να γίνει διαβούλευση. Βάσει τη πράσινη βίβλου θα υποβάλουμε τι προτάσει μα στην ανακοίνωση με διαφορετικέ εναλλακτικέ και όταν έχει, γίνει, όταν έχει ολοκληρωθεί και η συζήτηση επί τη ανακοινώσεω θα υποβληθεί η τελική νομοθετική πρόταση. Πάντω κάποια στοιχεία για μένα είναι σαφή, δηλαδή ότι χρειάζονται στοιχεία προβολή, στοιχεία επικοινωνιακά ή διαφήμιση τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αγορά για την εσωτερική ίσως θα έπρεπε περισσότερο να δώσουμε έμφαση στα στοιχεία που μπορούμε να αποστείλουμε στο ευρύ κοινό, στον ιδιώτη καταναλωτή. Τι σημαίνει δηλαδή γεωργικό προϊόν, τρόφιμο ευρωπαϊκό, τι προσφέρει σε σχέση με τα εισαγόμενα, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω δηλαδή πρέπει ο καταναλωτής να έχει συνείδηση του ότι κάθε προϊόν που κατεβάζει από το ράφι του σούπερ έχει ε, μία αξία προσθέμενη τη δουλειά δηλαδή του γεωργού ο οποίος τηρεί και σέβεται προδιαγραφές στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε. Χρειάζομαστε επίσης μέσα για να προαγάγουμε τα μέσα, για να προβάλλουμε τα μέσα ελέγχου της ποιότητας. Έχουμε ένα σχέδιο νομοθετικό τώρα ε, που συζητούμε και πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Ε, μια συζήτηση δηλαδή έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτή, να έχουμε λύσει ώστε να μπορεί ο καταναλωτή να καταλάβει καλύτερα τι σημαίνει το ευρωπαϊκό. Επίση έχουμε προτάσει για τι τοπικέ αγορέ ή τι αγορέ που απευθύνονται στην ευρεία κατανάλωση. Για δε το διεθνέ πεδίο θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αναζητήσουμε μέσα τα οποία μας επιτρέπουν με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να κάνουμε προβολή πακέτων ευρωπαϊκών προϊόντων με συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα διαβήματα ή προσπάθειες. Για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις είμαστε σε αμυντική θέση σε ορισμένε περιπτώσει αλλά και σε επιθετική, γιατί υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία όμω δεν είναι παντότε επαρκώ γνωστά. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμη αυτή την εβδομάδα, μέχρι το τέλο τη εβδομάδα, εγώ μεταβαίνω προσωπικό στην Κίνα σε μία επίσκεψη θα κρατήσει σχεδόν ολόκληρη εβδομάδα, το μεγαλύτερο μέρο τη οποία θα αφιερωθεί στην προβολή των ποιοτικών ευρωπαϊκών προϊόντων. Θα με συνοδεύσουν επιχειρηματίες, ε, παραγωγή τη γεωργική αγορά που εκπροσωπούν σήματα ποιότητα, ώστε να τα καταστήσουμε γνωστά στην κινέζικη αγορά, που πιστεύω τα περιμένει, μέσα δηλαδή προβολής τα οποία ε, θα στηριχθούν στην ε, έμφαση στην ποιότητα των δικών μας προϊόντων. Πάνω σε αυτό μπορούμε να στηριχθούμε. Και βεβαίως αν χρειαστούν περισσότερα οικονομικά μέσα, γιατί εγώ θα προτείνω στο συλλογικό όργανο της Επιτροπής ένα μια καλύτερη πρικοδότηση, σημαντικότερη πρικοδότηση από ό,τι έχουμε τώρα, τουλάχιστον για την προβολή. Και αφού γίνει συζήτηση, θα δούμε και ποιο είναι το καταλληλότερο διοικητικό πλαίσιο για τη διαχείριση αυτών των μέσων και τη σχετική πρικοδότηση. Χωρί να περιπλέκονται πολύ τα πράγματα, χωρί να είναι πολύ περίπλοκη η γραφειοκρατικά διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και κατά τρόπο που να επιτρέπει κάθε δυνατότητα αξιοποίηση ε, τη προβολή αυτή, των δυνατοτήτων προβολή. Κάπου θα χρειάζονται και εξειδικευμένε γνώσει. Άρα, ίσω θα μπορούσαμε ενδεχομένω αυτέ τι ειδικεύσει, εξειδικεύσει να τι τοποθετήσουμε σε μια χωριστή ε, οργάνωση, σε ένα φορέο, φορέα ε, χωριστό. Θα δούμε με τις προτάσεις ε, που θα έχουμε να καταθέσουμε, θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε φυσικά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αφήνουμε ένα χρονικό περιθώριο. Για δε τη Μερκοσούρ, είμαστε σε φάση προετοιμασίας των προτάσεων για την πρόσφορά μας. Προσφορά η οποία θα έχει χωριστή κατηγορία για τα προϊόντα τα οποία εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα ευαίσθητα, φερπίν προϊόντα ε, κρέατος, το κρέας και τα προϊόντα του που θεωρούμε ευαίσθητο προϊόν. Επίσης, ε, προκαταβάλουμε λίγο πολύ τις προτάσεις της Ντόχα και έτσι εισάγουμε στην προσφορά που καταθέτουμε προς τις χώρες Μερκοσούρ ήδη τη διάσταση που αναμένεται ότι θα ε, λάβουν ή την ε, τροπή που αναμένεται ότι θα λάβουν διαπραγματεύσει Δόχα. Για να είμαστε έτοιμοι και εκεί. Επίσης, προτείνουμε μία ε, λύση με προσφορά που θα παρουσιάζει διαφοροποίηση, διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή ανάλογα με το προϊόν. Επίσης, οι επίτροποι Κένταλη και Ποτόσνικ, με τους οποίους θα συνεχίσω τη συζήτηση και τις διαπραγματεύσεις, ε, θα ε, ενισχύσουν τις προτάσεις μας μέσα από τη διαπραγμάτευση αυτή, ε, εντάσσοντας προδιαγραφές παραγωγής, προδιαγραφές ποιότητας, προδιαγραφές δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων επιπτώσεως της παραγωγής επί των φυσικών πόρων. Αυτά λοιπόν. Αυτά θα αναπτυχθούν στη συζήτηση με το Μερκοσούρ. Δεν έχει προσδοριστεί το χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή των προσφορών. Είμαστε ακόμα στη φάση των προκατακτικών ε, συνομιλιών. Αλλά εμεί από πλευρά μα ε, λίγο πολύ ε, οριστικοποιούμε την προσφορά που θα υποβάλουμε. Έχουμε κάνει και τι πρώτε μελέτε επιπτώσεων. Έχω ζητήσει από τι υπηρεσίε μου να διευκρινίσουν ορισμένα σημεία για να έχουμε πιο συγκεκριμένε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις ε, των συναλλαγών αυτών, των ελεύθερων συναλλαγών αυτών σε συγκεκριμένα τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά όχι μόνο τμήματα ή τομείς, αλλά και συγκεκριμένα σε περιφέρειες που ενδεχομένως να πληγούν περισσότερο από την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Για την, προβολή των προϊόντων μίλησα για την απλούστευση. Κύριε Νίκολσον, συμφωνώ απολύτως. Θα πρέπει όχι μόνο να εισάγονται στοιχεία, αλλά και όταν εισάγονται στοιχεία θα πρέπει αυτά να έχουν σαν αποτέλεσμα να αποδεικνύουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική που είναι μια δημόσια πολιτική παράγει δημόσιο αγαθό, παράγει δημόσιο όφελος. Γι' αυτό το λόγο και μόνο πρέπει να προσθέτει, να προσθέτει νέες διατάξεις και για κανέναν άλλον. Η δε ε, πρόταση για γεωργικές πρακτικέ που μπορούν να επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων υπάγεται στον πρώτο πυλώνα και γιατί το έχω εξηγήσει πολλέ φορέ, διότι πρέπει να εξηγούμε ότι οι, πολιτική, οι οι άριστες γεωργικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν θετικά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορούμε να το συσχετίσουμε, να το συνδέσουμε με τον πρώτο πυλώνα και μόνο. Με το δεύτερο πυλώνα είχαμε συστήσει και πριν και επί τη ευκαιρία της και όπου είχαν τοποθετηθεί οι περισσότεροι, για να μην οι πάντε, στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της κάθε περιφέρειας, ε, τοπική δηλαδή, τα τοπικά χαρακτηριστικά και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε επίσης. Αν έχουμε κάποιους υποχρεωτικούς, αν έχουμε ε, στοιχεία υποχρεωτικά για το δεύτερο πυλώνα, στοιχεία υποχρεωτικά που θα ισχύουν για ολόκληρη την Ευρώπη, ούτε την, την οικονομία κλίμακας θα έχουμε, ούτε θα μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση να παραγάγει καλύτερα προϊόντα. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε περιφέρεια, κάθε περιοχή, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες και τον τρόπο ελέγχου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει κάθε περιοχή τη ιδιαιτερότητές της στην παραγωγή. Γι' αυτό να ζητούμε τον καλύτερο και απλούστερο τρόπο επαλήθευσης αυτών των στοιχείων. Ταυτόχρονα, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική ε, ρυθμιστική παρέμβαση. παρέμβαση το συζήτησα και με τον Επίτροπο Ποτνός και, θα έρθει και εκείνος με τις δικές του ε, υπηρεσίες και, και τις δικές του προτάσεις περί απλούστευσης των ε, μέτρων προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες ε, που είναι όχι μόνο διοικητικές αλλά και γενικές ε, συνέπειες ε, για ολόκληρη την κοινωνία της διασταυρούμενης συμμόρφωσης. Κύριε Λάιον, είπατε ότι κρύβεται η Επιτροπή, ότι δρά εν κρυφό και παραβίστο. Δεν νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον έχω ποτέ αποφύγει συζήτηση για κάποια πρόταση. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ ούτε και στην ολομέλεια της, των συνεδριάσεων της Επιτροπής σας, της Επιτροπής Γεωργίας, ούτε και έχω ποτέ ε, αρνηθεί διμερείς συνομιλίες με κάποιους ε, συναδέλφους σας. Ε, ίσως να μην έχω δει τον κύριο Νίκολσον τόσο πολύ, αλλά δεν θυμάμαι να του αρνήθηκα ραντεβού όποτε μου το ζήτησε, τον κύριο Νίκολσον συγκεκριμένα. Και τώρα αν θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού, κύριο Νίκολσον, εν πάση περιπτώσει το σημειώνω. Και πάντως με τους λοιπούς συντονιστές των πολιτικών ομάδων έχω συνεργαστεί και να ξέρετε ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Λέτε ότι δεν προσφέρονται αρκετά στοιχεία επί των προτάσεων αυτών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες ομοθετικές της προτάσεις ε, και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσουν και οι θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς, οι υπηρεσίε της Γενικής Διεύθυνσης ε, Άγκρη πάντα τα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλατε ε, να σας προσφέρουν. Και αυτό πάντοτε συνεχίζεται. Είμαστε στη διάθεσή σας και έχουμε κάθε πρόθεση να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα ανοιχτή συνεργασίας. Απάντησε επίσης πιστεύω στον κύριο Φοντάνα. Είπατε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν κάνει προτάσεις για ε, προδιαγραφές ποιότητας προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω όμως ότι ο χώρος για την διατύπωση τέτοιου είδου προδιαγραφών είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε στο εσωτερικό μας να θεσπίσουμε μία σειρά καρόνων που θα επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή σε μια άλλη χώρα. Ίσως, μέσα από το πλαίσιο τη ε, Παγκοσμίου Οργάνωσης Εμπορίου ε, μπορούμε, αν και βέβαια είναι και αυτό πολύ δύσκολο γιατί σε εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις είναι δύσκολο να εισαχθούν στοιχεία μη εμπορικά. Εν πάση περιπτώσει όμω, ό,τι μπορώ εγώ θα το ε, κάνω προκειμένου και στις ε, γενικότερες αυτές εμπορικές συνομιλίες ε, να εισαχθούν τα γεωργικά θέματα. Και ο κύριος είναι και ο κύριος Νταλή, όπω ξέρετε, ρημνούν για την διαφύλαξη των διατάξεων σχετικών με την προστασία τη δημόσιας υγεία και τη προστασία του καταναλωτή. Και είναι αυτονόητο ότι αυτά τα πράγματα δεν θα λησμονηθούν στις ε, ε, συνομιλίε μας με τους εταίρου. Κύριε Ρούμπιξ... Ξέρω ότι δεν είναι ίσω τώρα η στιγμή να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το χρονοδιάγραμμα, αλλά αν κοιτάξετε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δώσω μια απάντηση, προτάσει για την κυριαρχική πολιτική για την περίοδο μετά το 2013, θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την υποβολή των προτάσεων με καλύτερη κατανομή ε, των άμεσων ενισχύσεων. Πιο δίκαιη κατανομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ντάτσαν Τσόλο Με αυτή την πρώτη απάντηση που μας έδωσε στη, στα ερωτήματα των συντονιστών πιστεύω ότι έχουν αποσαφινιστεί πολλά. Θα γίνει λόγος και για το χρονοδιάγραμμα ως προς την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Υπάρχουν 18 μιλητές, 18 εγγεγραμμένοι. Έπρεπε να είχαμε οργανωθεί καλύτερα. Λάτενφελτ tempo il più possibile ristretto. A cukorpiacon kialakult feszültségről szeretném önt kérdezni. Az elmúlt időszakban jelent... Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. να ρωτήσω ένα θέμα σχετικό με την ε, οργάνωση, με την αγορά της ζάχαρης. Ξέρετε ότι έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα πολύ η, αγορά, η τιμή της ε, ζάχαρης. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα πρέπει κάπως να διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση, να αντιμετωπιστεί και ρωτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει δυνατότητα για αξιοποίηση ισογλυκόζης που προέρχεται από το καλαμπόκι. Αν μπορεί δηλαδή αυτή να διατεθεί στην αγορά. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν ε, εργοστάσια με πολύ με υψηλό δυναμικό παραγωγής. Ωστόσο η Επιτροπή ξέρουμε ότι είχε απορρίψει ανεφετέρω την ε, πρόταση και ως εκ τούτου παρεμποδίζει και την ανάπτυξη πολλών εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζει επίσης την ανάπτυξη νέων ε, νέου οικονομικού δυναμικού που μπορούν να προσφέρουν αυτές οι, αυτά τα εργοστάσια. Γιατί ξέρετε ότι αν ε, έχουμε τη δυνατότητα και, και προσφορά στην αγορά ισογλυκόζης από καλαμπόκι, ε, θα διπλασιαστεί ουσιαστικά η αξία του προϊόντος αυτού. Mm. Νομίζω ότι θα βοηθούσε αν δινόταν η άδεια και να μειωθούν τα ελλείμματα και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ε, πολύ ψηλής τιμής ε, ε, ζάχαρης. Δηλαδή ουσιαστικά εμποδίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προσφορά ζάχαρη σε οικονομική τιμή, γλυκαντικού σε οικονομική τιμή για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με το πνεύμα των προτάσεων για την Ευρώπη του 2020. Και θέσει εργασία δεν επιτρέπεται να δημιουργηθούν και παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα κάπτεται με την στάση αυτή και μειώνεται την ε, δυνατότητα για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ερωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, είστε διατεθειμένος να βοηθήσετε με τις επιλογές Ευρωπαϊκής Επιτροπής την εξυπηρέτηση των στόχων του 2020. Είστε διατεθειμένος να επιτρέψετε την λειτουργία αυτών των εργοστασίων παραγωγής της ή προτιμάτε μόνο να υποστηρίξετε τις εισαγωγές, κύριος Τσόλος. Κοιτάξτε, να απαντήσω αμέσως, μου επιτρέπετε. Από αυτά που λέτε είναι σαν να είναι η Επιτροπή ο, η πηγή κάθε κακού. Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να εφαρμόσει τις αποφάσεις του νομοθέτη, νομοθετικού οργάνου και Συμβουλίου, νομοθετικού οργάνου, δηλαδή Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Κάναμε ό,τι μα επέτρεπαν οι αγορέ σε σχέση με τη ζάχαρη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα προμήθεια, πάντα σε σεβασμό τη νομοθεσία. Δεν αποφασίζει απευθεία για τι επενδύσει στην ισογλυκόζη, σε οτιδήποτε άλλο, ζαχαρότευτλο, ζάχαρη ακατέργαστη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αποφασίζει η Επιτροπή τι είδου θέσει εργασία θα διαφυλάξουν οι μη επιχειρήσει οι οποίε απολύουν κόσμο. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν οι επιχειρήσει όταν απολύουν του εργάτε του. Και η Επιτροπή στι προτάσει τη κάνει ό,τι μπορεί λαμβάνοντα υπόψη ότι πρέπει και να διαφυλάξει την απρόσκοπτη λειτουργία τη αγορά τη ζάχαρη. Εγώ πάντα είχα ανοιχτό πνεύμα για συζητήσει, επιλογέ καινούριε για την αγορά τη ζάχαρη. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια ζάχαρη ε, βαρύτατα ρυθμιζόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστώσει και με τιμέ. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θα μπορούσε ή ό,τι θα ήθελε ή εν ό,τι θα μπορούσε να κάνει μια επιχείρηση αν ληφθεί, αν η απόφαση να καταργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς, η διαχείριση των αγορών, τότε θα πρέπει η κάθε επιχειρήση να αναλάβει τις ευθύνες της. Μέχρι τότε είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες των οικονομικών τους αποφάσεων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Θα χρειαστούμε 10 λεπτά περισσότερα από τον ε, Επίτροπο Γκαρσία, Ρέιμερς, σας παρακαλώ ε, ένα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Άκουσα να λέει ο κύριος Τσόλος ότι θα προωθήσουμε, θα, θα μας απασχολήσει η προώθηση προϊόντων. Αυτό το υπερασπίζομαι εδώ και πολλά χρόνια όμως ε, δεν χρησιμοποιείται σωστά το σύστημα πρόθεσης προϊόντων. Υπάρχουν ελλείμματα και διακρίσεις μεταξύ προϊόντων. Δηλαδή, ο ίνος δεν μπορεί να προωθηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό έτσι ώστε είναι πιο ευέλικτος ο μηχανισμός αυτός και για να μην γίνονται διακρίσεις όπως ισχύει στην περίπτωση του Ίνου. Αυτό θα ήταν λογικό και απολύτως απαραίτητο, διότι έτσι θα μπορέσει να γίνει εμπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των προϊόντων χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση γίνεται μεγάλη διάκριση κατά του κρασιού. Επίσης, για να μπορεί κανείς να προωθήσει την κοινοτική παραγωγή έναντι τρίτων χωρών θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαιότητα. Εάν δεν απαιτήσουμε από τις τρίτες χώρες που στέλνουν τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν απαιτήσουμε να υπάρχει ε, αλληλεγγύη, τότε δεν θα μπορέσει να ισχύσει ένα σύστημα αμοιβαιότητας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα γιατί διαφορετικά καμία ε, ρήτρα ασφάλειας δεν θα μπορέσει να ισχύσει. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα ελέγχων στα σύνορα να είναι αποτελεσματικό. Αυτό ισχύει στις ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά μαθήματα από εκεί. Επειδή δεν θα μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σήμερα, μπορείτε να μας πείτε πώς, θα, προωθούνται οι συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας σε σχέση με αυτές τις τροποποίησεις Ρέιμερς και μετά Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπουμε τακτικά για συζήτηση, για συνομιλία εδώ στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι για την παρουσίαση αυτή της προτάσεως για το πρόγραμμα εργασίας 2012. Βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα και της μεταρρύθμισης και της πολιτικής και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που παραμένουν εκκρεμή. Πάντω είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι λέτε ότι θέλετε με βάση δημόσια ακρόαση να αναπτύξετε την πράσινη βίβλο. Θα ήθελα να δω πώ θα γίνει αυτό βέβαια, γιατί στη δημόσια ακρόαση, στο δημόσιο διάλογο, διαβούλευση, ε, συνήθω επικρατούν κάποια ε, συμφέροντα. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δηλαδή εξισορρόπηση συμφερόντων και θέσεων και ο κλασικό γεωργό, η κτηνοτρόφος δεν μπορεί να κάνει να ξακουστεί η φωνή του. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε αυτό και επίση πώ θα προσδιορίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει μια ευελιξία ω προ την ε, παραγωγή, τη γεωργική αλλά και για, την, ε, για τον ίδιο τον παραγωγό, σε ποιο βαθμό δηλαδή, θα έχει την ελευθερία των επιλογών του και επίση για τι εμπορικέ συναλλαγές συχνά τίνουμε να επικεντρωνόμαστε πιστωρώ σε αυτά τα πράγματα που μας φοβίζουν. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θεωρώ θετικό το ότι εσείς προτιμάτε να στραφείτε προς ε, την ε, εξέταση περισσότερο των ευκαιριών που μας προσφέρονται. Πώς μπορούμε δηλαδή να προαγάγουμε τα προϊόντα μας, γιατί είναι καλύτερα, γιατί είναι ασφαλέστερα, γιατί μπορούμε να τα ε, διαθέσουμε σε όλο τον κόσμο. Και επίση μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε όχι το ψάρι, αλλά τον ψαρά, δηλαδή τον, ε, ε, τον καταναλωτή και όχι τον παραγωγό ότι είναι καλά τα προϊόντα. Ο τίτλος ήταν το πρόγραμμα εργασίας το 2012. Την πρώτη μέρα του 2012 θα αντιμετωπίσετε ένα μεγάλο πρόβλημα. 80 εκατομμύρια 80 εκατομμύρια αυγών θα παράγονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ναι. θα πρέπει να σε απασχολήσει διότι η παραγωγή αυγών αφορά όλη ολόκληρη την Ευρώπη και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι Βρετανοί παραγωγή δαπάνησαν 400 εκατομμύρια για να συμμορφωθούν, συμμορφωθούν με τον κανονισμό σας. Συνεπώς δεν μπορούμε να δεχόμαστε άλλοι να παράγουν παράνομα. Θα ήθελα μάλλον είδα ποιες ε, είναι οι εκμεταλλεύσεις, διότι όπως ξέρετε οι τιμές ε, των κλοβών ε, έχουν αυξηθεί και θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί το 2012. Μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό και να προωθείτε αυτά τα 80 εκατομμύρια αυγά με μία νεκροκεφαλή πάνω για να ξέρουμε ποιος, τι, ποιος τα παράγει και γιατί. Σε Κυριέσκη και μετά Μποβέ. Κύριε Επίτροπε, πότε ακριβώς θα μας υποβάλλετε τις νομοθετικές σας, την νομοθετική σας δέσμη. Ο κύριος Λεβαντόφσκι τον Ιούνιο φαντάζομαι θα υποβάλει το έγγραφό του και μετά θα χρειαστούν ίσως πέντε μήνες για να μεταφραστεί αυτό σε νομοθετήματα, αλλά αυτό είναι πολύ αργά πια. Αν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτρόπων, δεν θα μπορούσε από τότε που ο κύριος Λεβαντόφσκι θα έχει γράψει κάτι να γίνουν πιο γρήγορα τα νομοθετήματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσετε. Γιατί συμβαίνουν τέτοιες καθυστερήσεις και κάτι άλλο ακόμη. Το θέμα της καινοτομίας στη γεωργία και αυτό να το προσέξουμε περισσότερο στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και ένα τρίτο το βιωτικό επίπεδο και η ανέχεια στην Ήπεθρο καθώς και ο στρατηγικός συντονισμός που χρειάζεται. Θα συνεχίσετε να επιμένετε επί του συντονισμού ή το αφήσατε πια αυτό. Ευχαριστούμε Μπόβε και μετά Ντόρφμαν. Επίτροπε, αρχίζω λέγοντας ότι ανησυχώ για την πίεση που ασκούν πέντε κράτη τουλάχιστον που λένε ότι αρνούνται τα ανώτατα όρια που έχετε προτείνει στις επιχορηγήσεις. Ανησυχώ λοιπόν για τις πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες αγροβιομηχανίες που και η παραγωγή ζυζανιοκατώνων και παρασιτοκτώνων. Αν θέλετε να μειωθούν τα καλακτοκομικά σε 30% άλλοι δεν λένε αρκούν τα 20% τι θα γίνει. Δεν πώς θα ελέγξουμε τις τιμές. Έπειτα ανησυχώ επίσης και επανέρχομαι εδώ στο θέμα της ποιότητας για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τις ελεύθερες συναλλαγές πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η προώθηση μέσα στην Ευρώπη των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων εάν ταυτόχρονα το κόστος είναι απαγορευτικό και για το βόλιο κρέας αλλά και για τα δαμάσκηνα που τους επιτίθενται οι αγορές αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Οι κανόνες που μας επιβάλλονται θεωρούν πάντοτε τη γεωργία ως κάτι ανταλλάξιμο με τον τομέα των υπηρεσιών. Όχι. Εμείς δεν δεχόμαστε πια αυτόν τον ρόλο για τους γεωργούς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Ζωζέ. Ο Ντόρφμαν και μετά Μάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην ε, πράσινη βιβλό. Πολύ καλό το ότι σκοπεύετε να υποβάλετε μία πρόταση ε, για τις ε, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε πρόβλημα ως προς την, τα ποσοστά επί των συνολικών γεωργικών δαπανών που έχουμε για, την, ε, για τις δαπάνες αυτές που είναι χιλιοστό μόνο επί των γεωργικών ε, δαπανών και δεύτερον ως προς το περιεχόμενο Μπορεί να λέτε ότι θα γίνει προβολή των γεωργικών προϊόντων. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με προϊόντα ε, βιομηχανικά, προϊόντα τα οποία ε, ε, φτάνουν μέχρι τα ράφια του σούπερ μάρκετ, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για συγκεκριμένη προβολή. Γιατί είναι πολύ λιγότερο διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να μπουν πάνω σε αυτό, να ανέβουν πάνω σε αυτό το τρένο και να ανοίξουν το πορτοφόλι για συγχρηματοδότηση. Πολύ καλό το ότι θα επισκεφτείτε την ε, Κίνα. Φαντάζομαι ότι θα κοιτάξετε περισσότερο να προβάλλετε τα προϊόντα τα οποία έχουν ε, και κάποια ένδειξη προελεύσεως, αυτά τα οποία μπορούν να πουληθούν καλύτερα δηλαδή. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προφυλάξουμε και τις δικές μας αγορές από αντίστροφε ροές προϊόντων. Επίσης, το Κοινοβούλιο το Μάιο κατέθεσε μία πρόταση για τις απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές. Μετά από αυτό η Επιτροπή δεν αντέδρασε καθόλου. Δεν ακούσαμε τίποτα από πλευρά τη Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι έχει γίνει αυτή η υπόθεση στο δικό σα επίπεδο. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις εντάχει. Σε σχέση με τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, μιλήσαμε για τις χώρες Μερκοσούρ καταρχήν. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο υπάρχουν προβλέψεις μέχρι το 2012 να υπάρξουν νέες συμφωνίες στον αγροτικό γεωργικό τομέα. Ε, μέσα στα πλαίσια του χωρών όπως το Εκουαδόρ που έχει υψηλή, υψηλό ποσοστό καλλιέργειας ε, μπανάνας. Επίσης με το Μαρόκο γίνεται μία συζήτηση σε σχέση με αυτή τη συμφωνία που υφίσταται και υπάρχει πρόταση να απορριφθεί, διότι υπάρχουν ε, θέματα ποσοστώσεων και τιμών που δεν έχουν συμφωνηθεί και υπάρχει και το θέμα των ελέγχων. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο στο εγγύς μέλλον, όπως σας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αλλάξει ο κανονισμός τιμών αναφοράς οποροκυπευτικών και επίσης ως προς την παραγωγή ντομάτας του, από πλευράς Μαρόκου, βασιλείου του Μαρόκου, υπάρχουν ε, μεγάλες ε, μεγάλες αντιφάσεις διότι για 25 μέρες έγινε πώληση ε, τομάτας η οποία δεν ανταποκρινόταν στις ε, τιμές κόστους. Επίσης, τι θα γίνει με την καλλιέργεια μπανάνας. Θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Επίτροπος να αλλάξει την αξιολόγηση, να δούμε τι επιπτώσεις ε, υπάρχουν σε σχέση με τη μείωση των ποσοστώσεων. Θα ήθελα να μην μιλήσουμε το 2012 πλέον για το θέμα της μπανάνας. Γεια. Και μετά Γκαρσία πέρασε. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι πάντα στη θέση μα στην Επιτροπή για συζήτηση. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καταστεί σαφέ και το οποίο έχει θίξει κάποιου συνάδελφου ήδη. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την πρόταση που αναφέρατε ότι οι νομοθετικέ προτάσει θα δημοσιευθούν όταν είναι στη θέση σα και οι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Πολύ καλά. Αυτό όμω αντίστροφα. Μήπω σημαίνει ότι οι δημοσιονομικέ προοπτικέ προκειμένου να. Ε, προετοιμαστούν, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν τι γεωργικές προτάσεις αντίστροφα. Δηλαδή πω καθυστερήσουν οι δημοσιονομικές προοπτικέ σε αναμονή της υποβολή των δικών σα προτάσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευράς Επιτρόπου έγινε λόγος για το ποιοτικό πακέτο και θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να γίνουν αλλαγές. Θα γίνει ένα σεμινάριο σήμερα το απόγευμα από όσο γνωρίζω και πιστεύω εντάχει να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε οπωσδήποτε. Τη στιγμή που θα υπάρχει αυτό το πακέτο, το θέμα που προέχει είναι η προώθηση. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς επειδή θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει η στρατηγική μας, θα πρέπει να είναι ευέλικτη, αποτελεσματική και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα κοινοτικά προϊόντα είναι γνωστά και προς τα έξω. Γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με ευελιξία και σπουδή. Στεφάν Λεφόλ και μετά Παπαστάμκος. Ναι, σύντομα γιατί πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Το πρόγραμμα το είχαμε δεχτεί από το για, το για το φθινόπωρο. Αλλά η ποιότητα πρώτον, πολύ σημαντικό στοιχείο, πρέπει να προσέξουμε. Σήμερα υπάρχει θέληση μείωσης της ισχύω της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, δηλαδή της ποιότητάς της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το γάλα και εκεί θα υποβάλω τροπολογίες. Υπάρχει κίνδυνο, σας το λέω ανοιχτά και παρακαλώ την Κομισιόν να το προσέξει ιδιαίτερα. Και από τον ΠΟΕ γίνονται αυτές οι επιθέσεις και από αλλού. Το γαλακτο, τα γαλακτοκομικά με την ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τώρα. Για τη μεταρρύθμιση και την σχετική έκθεση. Εγώ συμμερίζομαι τις απόψεις σας κύριε Επίτροπε. Πρέπει η γραμμή που θα ακολουθήσουμε να είναι ευνόητη, όχι να είναι συνεχώς οι και πότε από εδώ, πότε από εκεί. Πρέπει γι' αυτό να γίνει κάποτε μια ειλικρινή συζήτηση που θα μπορούσε ήδη να είχε γίνει πριν κατατεθούν οι τροπολογίες, αλλά θέλω μια σαφή γραμμή, ώστε μετά στη νομοθετική δέσμη να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και εκπλήξεις. Ευχαριστούμε Στεφάν Παπαστάμκος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την ανταπόκρισή του σε αυτή την διαθεσμική συνεργασία και θέλω να πω ότι προσωπικά δεν τον κατατάσω στους υπερόπτες επιτρόπους αλλά στους συνεργάσιμους ε, επιτρόπους γιατί υπάρχουν και υπερόπτες επίτροποι. Ε, κύριε Πίτροπε, αναφερθήκατε στο impact assessment και στη σχέση με την συμφωνία, τη συμφωνία με Μερκοσούρ. Εμεί, την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεσή μου με θέμα διεθνέ Ευρωπαϊκή Γεωργία και Διεθνέ Εμπόριο και εκεί υπάρχει ρητή αναφορά ότι το impact assessment πρέπει να δημοσιοποιείται πριν από την ανταλλαγή προσφορών, πριν από το exchange of offers, είτε με τη Mercosur αύριο θα έχουμε την, τον Καναδά, έχουμε την Ινδία. Και επειδή δείχνεται ευαισθησία απέναντι στην κοινοβουλευτική βούληση, θα το λάβετε αυτό υπόψη. Και γνωρίζετε πολύ καλά, δεν μπορείτε να προκαταλάβετε την έκβαση των διαπραγματεύσεων του γύρου της Δόχα και εκεί το mandate, το διαπραγματευτικό, κάνει ρητή διασύνδεση ε, της έκβασης αυτής με τις, ε, των διαπραγματεύσεων με τις χώρες ε, της, ε, της Μερκοσούρ. Και μια κουβέντα ακόμα, Αναφερθήκατε στη ζάχαρη. Ναι, δεν νομοθέτησε η Κομισιόν. Η Κομισιόν πρότεινε, αλλά ήταν επιμονή της προκατόχουσα στην Κομισιόν, η οποία οδήγησε και της ορθοδοξίας τη γραφειοκρατία τη Κομισιόν, η οποία οδήγησε σε κλείσιμο εργοστασίων, σε απώλεια θέσεων εργασία, ήταν οι προτάσει τη Κομισιόν που κατέστησαν τη Βραζιλία ηγέτιδα δύναμη στον τομέα τη ζάχαρη και μεταφέρθηκαν συμφέροντα όχι υπέρ των αγροτών εκεί, αλλά υπέρ ολιγοπολιακών καταστάσεων. Και αυτό δεν τιμά ούτε την Κομισιόν, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ως προς τη νομοθετική πρόταση, ε, θα θέλαμε ως προς την αναθεώρηση της ΚΑΠ, ελπίζουμε να έχουμε την πρόταση νωρίς το φθινόπωρο και όχι προς το χειμώνα. Βεβαίω θα συζητήσουμε τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα του προϋπολογισμού, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι οι προτάσεις σας σε σχέση με την πρόθεση προϊόντων, ε, προώθηση εμπορικού σήματος και ποιότητα τροφίμων. Αυτές είναι πολύ, αυτή είναι πολύ σημαντική τομή και χαίρομαι για τις προτάσεις σας. Αν θέλετε να υποστηρίξετε τους αγρότες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, τότε ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος πυλώνας θα επιλύσουν τα προβλήματα, αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κατάσταση θα επιληθεί μόνο αν μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, που είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν έχουν μια καλή τιμή. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα κατασπαταλήσουμε δυνάμεις και πόρους. Θα αλλάξουμε λοιπόν τη διάρθρωση της παραγωγής και βεβαίως θα ε, βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής των αγορατών. Γι' αυτό θα ήθελα περαιτέρω στοιχεία από εσάς σε σχέση με αυτούς τους τομείς που προανέφερα. Δηλαδή καταρχήν η ποιότητα και η πρόθεση προϊόντου. Μισελ Νταντέν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για την διάθεση για συνομιλία. Βεβαίω, έχουμε το μάτι στραμμένο προ το μέλλον και τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και το παρελθόν και τι υπόλοιπε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα και δεν μπορούμε να αφήσουμε την αγορά να ρυθμίσει τα πάντα και να διαπιστώσουμε στη συνέχεια ποιε ήταν οι ζημιές που υπέστημεν. Σήμερα και μάλιστα το είχε πει και το Κοινοβούλιο στην, σε ένα ψηφισμά του, ο τομέα τη της αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο, ενώ ο τομέα τυρών σιτηρών τα πάει πολύ καλά, ίσω και παραπάνω από καλά. Έτσι λοιπόν ρωτώ, θα πρέπει το 2014 να περιμένουμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τόσο πολύ. Τιμέ των εισιτηρών αυτή τη στιγμή έχουν σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν να ακούγονται κάποιες φήμες ότι που κυκλοφορούν εδώ στα κτίρια μας ότι δεν χρειάζονται πια οι ε, στηρίξει στην ε, γεωργία και ο γεωργικός προϋπολογισμός εν γέννη μπορεί να λησμονηθεί. 300 ευρώ για τον τόνο ή 600 ε, για το εκτάριο παρά είναι πολλά ποσά. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να μετακυλήσουμε το, την έμφαση και να κοιτάξουμε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη γιατί σαν τις μύγες που οι επιχειρήσεις στην γεωργία μας, στην κτηνοτροφία μας καλύτερα δεν υπάρχει δυνατότητα για τον κτηνοτρόφο να εξασφαλίσει το εισόδημά του. Εμείς κοιτάμε δε αμέριμνα στο μέλλον και ατενίζουμε. Νομίζω τώρα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις που αφορούν το παρόν, που, κύριε Επίτροπε, ε, αποφάσεις που ταυτόχρονα θα δώσουν και ένα σαφέστατο μήνυμα για τον παραγωγό, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον ασχολείται με τα θέματα του προπολογισμού στο κοινό βουλίο. Και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας. Πρέπει να δώσουμε τον τόνο εγκαίρος και μάλιστα τη στιγμή που είναι τόσο υψηλές τιμές των σιτερών. Ευχαριστώ, Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Έχουμε εκκρεμότητα ακόμη και στην κοινή οργάνωση αγοράς για τα αμπελοϊνικά προϊόντα που κανονικά έχει οριστεί ως ορίζοντα το 2015. Ωστόσο, ε, έχει δοθεί μία υπόσχεση περί επανεξέτασης των προτάσεων αυτών το 2012. Έχετε κάνει κάτι, θα μας υποβάλλετε τη σχετική έκθεση, την ενδιάμεση έκθεση γιατί έχουμε παλαιότερες εκθέσεις και μελέτες του 2004 από πια δεν είναι χρήσιμες. Έχουν επισέλθει το μεταξύ αλλαγές και στην κοινή οργάνωση αγοράς ε, που έχουν να κάνουν και με την κατάργηση της ε, ε, διακοπής της παραγωγής, έχουμε να κάνουμε με διάφορες νέες λύσεις τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουμε μέσα από μια ενδιάμεση έκθεση για να δούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. ο αμπελοπαραγωγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζει ότι θα μπορέσει να επιβιώσει και μετά το 2014. Αυτό μου λένε διαρκώς οι παραγωγοί, οι δικοί μου της δικής μου περιοχή τουλάχιστον, να αγωνιούν για το μέλλον τους και την επιβίωσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Πατράω Κύριε Επίτροπε, Μία από τις, ε, από τα μεγαλύτερα μου, ένα από τα μεγαλύτερα μου ελλείμματα είναι το πακέτο προϊόντων γάλακτος και βλέπω ότι ως προς το δίκτυο διανομής δεν υπάρχουν ε, αλλαγές. Διότι έτσι όπως είναι ακροτηριασμένο το πακέτο γάλακτος δεν θα μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα που προτίθεται να επιλύσει σε σχέση με την εξαιρετική πρωτοβουλία που μας υποβλήθηκε για την ε, προώθηση των αγροτικών προϊόντων, υπάρχει ένα παράλληλο πρόβλημα. Η Επιτροπή Γεωργικών Προϊόντων θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλες επιτροπές ιδιαίτερα για την προστασία και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν ξέρω κατά πόσο στο εγγύης μέλλον για το πακέτο γάλακτος και για την διατροφική ασφάλεια θα μπορέσουμε να προωθήσουμε πραγματικές αγροτικές ε, πολιτικές που να έχουν όμως έναν εγκάρσιο χαρακτήρα. Επίσης, σε σχέση με το ΠΟΣΕΙ, το οποίο συζητιέται τώρα, θα ήθελα να τονίσω ότι το ΠΟΣΕΙ είναι ο μόνος μηχανισμός που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες έτσι ώστε να έχουν επαφή με την υπηρετική Ευρώπη και θα ήθελα να, δώσετε, να προσδώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ. Κανιέται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να, επιτρέψω, να επιστρέψω στο θέμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που είναι από τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους Ευρωπαίους γεωργούς. Το πρόγραμμά σας, στο πρόγραμμά σας θα ήθελα να ρωτήσω τι θεωρείτε μεταβατική περίοδο, πόσο θα διαρκέσει, γιατί ακούγονται διάφορες προτάσεις. 2020, 2025... Η προηγούμενη μεταρρύθμιση χρειάστηκε τέσσερα χρόνια μεταβατική περίοδο. Θα ήθελα να ξανασκεφτούμε την πιθανότητα οι χώρες μέλη που στην τωρινή περίοδο είχαν λάβει επιχορηγήσεις κάτω του μέσου όρου της Ένωσης να έχουν μικρότερη μεταβατική περίοδο. Και τώρα τα αντικειμενικά κριτήρια της μεταρρύθμισης. Στην έκθεση Lion που είχε εγκριθεί πέρυσι, συγχωμοφωνήσαμε όλοι και όλες ότι οι άμεσες πληρωμές πρέπει να γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια. Σας ζητώ λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η θέση σας για τα αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν το λόγο. Έγινε εδώ question time εδώ μέσα με τον Επίτροπο. Λοιπόν, και τώρα αυτός ο τελευταίος θα απαντήσει και με τις απαντήσεις του Επιτρόπου λίγη η συνεδρίαση θα ξαναρχίσει στις 3. Ορίστε κύριε Τσόλος μου. για τις προωθήσεις. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά που έχω ήδη πει. Σας είπα είναι ακόμη σχέδιο. Το επεξεργαζόμαστε ακόμη. Θα έχετε την πράσινη βίβλο και την ανακοίνωση πριν γίνουν οι νομοθετικές προτάσεις. αφού σας λέω είναι κάτι που το ετοιμάζουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες αφού δεν τις έχουμε επεξεργαστεί. Όταν θα είναι έτοιμες θα σας τις πούμε. Βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας την ιδιαιτερότητα ορισμένων τομέων, ορισμένων προϊόντων, το κρασί, τα λαχανικά, τα οποροκή πεφουτικά. Θα δούμε αν πρέπει να καταργηθούν ή όχι μερικές επιχορηγήσεις, θα δούμε ποιες λειτουργούν, ποιες όχι, πώς. Γενικά τις ιδιαιτερότητες, ώστε να έχουμε μία συνοπτική και συνεπή προσέγγιση Όποτε υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τομείς που λειτουργούν πολύ καλά δεν θα τις καταστρέψουμε, είναι προφανές. Λοιπόν τώρα για... για... όχι για... Κάθε φορά που θέτουμε ένα θέμα επανέρχεστε εσείς στο θέμα της αμοιβαιότητας και των ελέγχων στα σύνορα. Αλλά το ότι πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και μια πιο επιθετική προσέγγιση όταν χρειάζεται. Θα βρούμε τα εργαλεία για την καταλληλότερη πρόθεση. Για τους ελέγχους στα σύνορα σας έχω ξαναπεί επίσης ότι υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική για τον έλεγχο στα σύνορα που την εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, αρμόδιες υπηρεσίες των το θέμα δεν είναι πώ θα υπάρξει καλύτερη νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Το θέμα είναι να εφαρμόζεται. Και αν δεν εφαρμόζεται σωστά, δεν πταίει ούτε το Κοινοβούλιο ούτε η Κομισιόν. Πρέπει να το δούμε και αυτό. πώ οι Ισπανικές, Ιταλικές αρχές και άλλες, ας μην τα αναφέρω όλα τα κράτη, έχουν προβλήματα. Αυτές οι αρχές όμως πρέπει να τα λύσουν. Τώρα, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Δεν θέλω να γίνω εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ μέσα. Αν θέλετε, καλέστε τον Ουγγροϊπουργό ή και τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα σας πει πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Και εγώ περιμένω να ακούσω. Την Πέμπτη θα δούμε τι θα πει το Συμβούλιο για τα συμπεράσματα επί της ανακοίνωσης της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση. Αλλά τι άλλο να σας πω. Εγώ δεν πήγα στις προκαρασκευαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Κυρία Ρέινερ, με την πράσινη βίβλο και μετά με την ανακοίνωσή μας θα δοθούν αυτές οι δύο τουλάχιστον ευκαιρίες για να συμμετάσχετε όπως πρέπει στη συζήτηση της πρότασης αυτής για την πρόθεση. Και την προετοιμασία αυτή την κάνουμε ακριβώς για να μπορέσει να υπάρξει συζήτηση. Πρώτα η πράσινη βίβλος και μετά η ανακοίνωση. Εγώ δεν βλέπω για τα αυγά να χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο χωριστό. Θα συμπεριληφθούν και τα αυγά στην πρόταση προώθησης. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Η πολιτική αυτή της προώθησης δεν στοχεύει ιδιαίτερα έναν τομέα περισσότερο από άλλους. κύριε Όχι, δεν χρειάζομαι πέντε μήνες για να χωνέψω τις ιδέες του Γιάννου Λεβαντόφσκι. Οι ιδέες αυτές υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι γιατί η Κομισιόν πρέπει να μπορέσει να τελειώσει την μελέτη αξιολόγησης και τη διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτή δεν μπορούμε να την κάνουμε πριν ακουστούν οι προτάσεις του προϋπολογισμού. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά η χρονική. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που δεν μπορούμε να τις συντομεύσουμε. Για την καινοτομία στη Γεωργία, ναι, είναι ένα θέμα που όπως είπα επανειλημμένα θα το ξαναπούμε πολλές φορές όσο για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα δοθούν ευκαιρίες ειδικά. Δεν χρειάζεται όμως να μετατραπεί η ΚΑΠ απλώς σε κοινωνική πολιτική. Θα έχει όμως κοινωνικά στοιχεία, είναι προφανές. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να κάνουμε τον απαραίτητο συντονισμό. Κύριε Μποβέ, πώς θα προωθήσουμε προϊόντα εφόσον υπάρχουν επιθέσεις με εισαγωγές, κοιτάξτε. Η πολιτική αυτή δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα μεν, αλλά νομίζω ότι οι καταναλωτές και καταναλώτριές μας θα γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών και μη προϊόντων. Είναι κάτι που θα έπρεπε νομίζω να γίνει, που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αν υπάρχουν φραγμοί που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, τουλάχιστον να υπάρξει η πληροφόρηση ώστε η επιλογή του καταναλωτή και της καταναλώτριας να είναι πιο ακριβής. Πρέπει όμως να γίνει μια πρόθεση των ευρωπαϊκών προϊόντων για να γνωρίζουν όλοι ποιες είναι οι διαφορές με τα άλλα. Κύριε Ντόρφμαν, νομίζω ότι απάντησα επίσης στα ερωτήματά σας, τουλάχιστον μερικά. Αλλά αν δεν τις απάντησα όλες είναι γιατί ακόμη τις επεξεργαζόμαστε ορισμένες πτυχές. Δεν εννοώ πάντως ότι δεν θα λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων, τα κρασιά κτλ. Έχουμε και χωριστά εργαλεία για τα απορροκυπευτικά και λαχανικά. Υπάρχουν οι διαβουλεύσεις μας με τις οργανώσεις των παραγωγών. Μπορούμε όμως ίσως να βρούμε και άλλα πρόσθετα στοιχεία που να προσαρμοστούν και για άλλους τομείς και να υποφεληθούν και τα προκυπευτικά και τα κράσια από αυτό. οι ιδιαιτερότητες που αφορούν προϊόντα ιδιαίτερα σημαντικά για την υγεία των καταναλωτών και καταναλωτριών θα ληφθούν επίσης υπόψη για το κρασί. Ας πούμε δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά μπορούμε να κάνουμε μία πρόσθετη προώθηση, χωρίς να παραβιάσουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα κάνω εγώ την αλλαγή. Αν θέλετε συζητήστε το με τον Επίτροπο Ντάλι τι επιπτώσεις έχουν τα διάφορα ποτά επί της υγείας των καταναλωτών και καταναλωτριών. Δεν μπορώ αυτό να το λύσω με ένα εργαλείο προώθησης ή διαφήμισης. Υπάρχουν ε, πάντως τα περιθώρια ελιγμών. Μην μου ζητάτε τα αδύνατα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τα αδύνατα. Έτσι είπα και εγώ απαντάει σε μία ερώτηση που δεν ακούστηκε. Αυτό ακριβώς μάλιστα είχα πει και εγώ. Αυτό. Να αυτό αυτό. Ακούστηκαν πολλά ερωτήματα για τη συμφωνία με το Μαρόκο και τον κανονισμό για τις ντομάτες και άλλα αποκλειστικά ως προς το Μαρόκο. Η μπάλα βρίσκεται στο δικό σας τμήμα του γηπέδου. Το ίδιο ισχύει και για άλλες νομοθετικές προτάσεις, για τα γαλακτοκομικά ας πούμε. Πάλι εσείς πρέπει να κάνετε το επόμενο βήμα. Η συμφωνία πάντως με το Μαρόκο προβλέπει μία συμφωνία με το Μαρόκο προβλέπει προστασία και οι εθνικές αρχές θα επιβάλλουν τους ελέγχους στα σύνορα μόνες τους. Δεν θα το κάνουν οι υπάλληλοι της Κομισιόν αυτό το πράγμα, τον έλεγχο στα σύνορα δηλαδή. Τα εργαλεία που έχουμε πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. πρόθεσή μου πάντως δεν είναι να γίνει κάποιος πόλεμος. Εγώ είμαι ειρηνικός άνθρωπος, θα το έχετε παρατηρήσει. Δεν έχω την πρόθεση ούτε να αρχίσω, ούτε να συνεχίσω πόλεμο, ούτε με για τις μπανάνες, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Η ΕΕ, πράγματι στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ πρέπει να υπάρξει και κάποιο συμπέρασμα για τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι προφανές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έληξε η νομοθετική διαδικασία αν δεν συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους. Αλλά επί πολλών συγκεκριμένων σημείων της μεταρρύθμισης μπορούμε να αποφασίσουμε τα πράγματα και την τελική απόφαση να την πάρουμε μόνον όταν θα έχουν κανονιστεί και τα δημοσιονομικά. Θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Μερκοσούρ και Παπαστάμκος. Για τα θέματα αυτά, πράγματι, δική μου ευθύνη είναι να προετοιμάσω αυτή την αξιολόγηση και την προσφορά, αλλά ο τρόπος παρουσίασης αυτών των πληροφοριών πρέπει να γίνει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν, γιατί δεν θα αφορούν όλα αυτά μόνον τον αγροτικό τομέα. Πρέπει να δούμε οι αξιολογήσεις πώς θα γίνουν στο σύνολο των τομέων που διαπραγματευόμαστε. Σημείωσα πάντως το αίτημά σας και θα προσπαθήσω να συντονιστώ με τον Ντεχούχτ. Για τη ζάχαρη το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν μιλάμε για τα αποτελέσματα του τομέα αυτού πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ευρωπαϊκός τομεύς της ζάχαρης ε, λειτουργεί καλά ή έχει ανταγωνιστικές τιμές. Και θα σκεφτούμε την μεταρρύθμιση του τομέα αυτού στα γενικότερα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ για να δούμε ποια θα ήταν τα καλύτερα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε ταυτόχρονα να πετύχουμε την προστασία του τομέα αλλά και να τους δώσουμε του δώσουμε την ευκαιρία να ωφεληθεί ανταγωνιστικά από τη διεθνή κατάσταση για να μην πάρει τη θέση της Ευρώπης η Βραζιλία ας πούμε. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και τη διαχείριση του τομέα διοικητικά και τη διεθνή αγορά. Κύριε Νταντάν τώρα. Είχα πει σε μια ολομέλεια ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας ως προς τις επιχορηγήσεις ενώ τις άμεσες παροχές. Για το χείριο και τα πουλερικά ξέρετε ποια εργαλεία διαθέτουμε. Όταν διαπραγματεύομαι με προσώπους των τομέων αυτών δεν άκουσα κανέναν να ζητάει πολύ πιο αυστηρή νομοθεσία ή τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν νομοθετικές προτάσεις που να επιταχύνουν τα πράγματα, γιατί υπάρχει ήδη το θέμα της συναπόφασης για την ΚΑΠ που απαιτεί μήνες ολόκληρους και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία διαθέτουμε. Χωρίς να παραβιάσουμε όμως ή όπως είπα και πριν τις δυνατότητες που πρέπει να έχει ο τομέας αυτός να ανταγωνιστεί διεθνώς. Για τα γαλακτοκομικά τα είπα. Εσείς θα κάνετε το επόμενο βήμα. Πρέπει να λάβει θέση το κάπα. Για το ΠΟΖΕΗ τώρα θα δούμε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά όταν τεθούν τα προβλήματα. Κυρία Κανέτες, για τη μεταβατική περίοδο. Δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει μεταβατική περίοδο που να ξεπερνάει την περίοδο Έγκριση ή ανάλυση του προπολογισμού ή χρήση του προπολογισμού. Αυτό δεν γίνεται, υπάρχει ένα όριο. Τώρα, τι ακριβώς περίοδο θα το συζητήσουμε όταν γίνουν οι νομοθετικέ προτάσεις. Με... Και θα δούμε με τι επιχειρήματα. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα συζητηθεί πολύ έντονα μεταξύ των τριών οργάνων. Όσο για τα αντικειμενικά κριτήρια, αναλύουμε την περίπτωση να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά κριτήρια, κάνουμε μία εξομοίωση. Δεν είναι εύκολο το θέμα γιατί δεν ξέρουμε αν και με τα αντικειμενικά κριτήρια δεν καταλήξουμε τελικά να χειροτερέψουμε τις ανισότητες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα κριτήρια και τι επιπτώσεις έχουν σε σχέση με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Αν θα υπάρξει περισσότερη σύγκληση αλλά και ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ της παραγωγής ενός σε σύγκριση με άλλο κράτος μέλος. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός εδώ μεταξύ αντικειμενικών κριτηρίων και περισσότερης σύγκλησης και μείωσης ανισοτήτων. Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε επίσης όταν επεξεργαστούμε τις νομοθετικές προτάσεις. Θα ακούσουμε τι έχετε να πείτε κι εσείς στις εκθέσεις που ετοιμάζεται. Αυτά. Ελπίζω να έχω απαντήσει, αν και ξεπέρασα λιγάκι το χρόνο μου, αλλά άλλη φορά μπορεί να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. σας υπενθυμίζω ότι στις 3 θα αρχίσουμε με το πακέτο γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας παρακαλώ να είστε ακριβείς στην ώρα σας για να μην χάσουμε το workshop.